Panie i Panowie, e, Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι μου. Κύριοι, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στη συνεδρία της Επιτροπής ε, ΣΕΔΕ, Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας. Νομίζω ότι έχετε πάρει όλοι τους φακέλους και έχετε και την ημέρα διάταξη κατά συνέπεια. Αυτό είναι το σχέδιο ημερησίας διάταξης για σήμερα και για αύριο. Εάν δεν υπάρξει κάποια αντίρρηση ή ένσταση σε σχέση με την ημερησία διάταξη, θα θεωρήσουμε ότι έχει εγκριθεί όσα έχει η ημερησία διάταξη. Πρέπει να σας ε, υπενθυμίσω ότι έχουμε και διερμηνία στις ε, γλώσσες όμως μόνο των πλήρων μελών της Επιτροπής μας. και η συνεδρίασή μας επίσης θα ε, εκπαιμφθεί και στο διαδίκτυο. Κάτι ακόμα που θέλω να σας αναφέρω είναι ότι ήμουνα στην Γεωργία, στην Τυφλίδα όπου παρακολούθησα μία συνδιάσκεψη σε σχέση με την ασφάλεια στο Νότιο Κάφκασο. Στα πλαίσια αυτής της επίσκεψης επίσης έχω συναντήσει την ε, υπηρεσία παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης, τον επικεφαλής λοιπόν και τα μέλη αυτής της Επιτροπής Παρακολούθησης. Υπάρχει λοιπόν και μία έκθεση πληρέστερη που μπορώ να σας διανύμω ή μάλλον που η γραμματεία μπορεί να σας διανύμει για το θέμα αυτό. Και επίσης επισκέφτηκα μια φυλακή όπου ήταν τρεις σημαντικοί πολιτικοί, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο πρώην Υπουργός Άμυνας της Γεωργίας και ο Δήμαρχος της Τυφλίδος. Και για το θέμα αυτό θα σας δώσω εν καιρό μια πλήρη αναφορά για τα θέματα αυτά. Έρχομαι λοιπόν στο σημείο ημερήσιας διάταξης, συνεχίζει η πρόοδος στα αγγλικά. Πρόκειται για τα θέματα κυβερνοασφάλειας και άμυνας. Έχουμε τρεις εξέχοντες ομιλητές στο πάνελ μας. Θα ήθελα καταρχήν να καλωσορίσω τον καθηγητή Ούντο Χέλμπρεχτ, ο οποίος είναι ο εκτελεστικός διευθυντής της ΕΝΙΣΑ, του Ευρωπαϊκού Φορέα για την Ασφάλεια των Δικτύων και της Πληροφορίας. Θα είναι ο πρώτος μας ομιλητής. <coughs> Ακολουθεί ο κ. Ρούντολφ Ρόι, ο οποίος είναι γνωστός, είναι ο διευθυντής ο αρμόδιος <coughs> για την πολιτική ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Και έχουμε και τον κύριο Πίτερ Ράουντ, ο οποίος είναι σμήναρχος από την ε, Βρετανική Γραφ και ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή διευθυντής στον Ευρωπαϊκό Φορέα Άμυνας. Το θέμα λοιπόν της ε, κυβερνοάμυνας και κυβερνοασφάλειας είναι ένα θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και θα είναι το αντικείμενο των παρουσιάσεων των καλεσμένων μας και είναι κάτι το πολύ σημαντικό εν ώψη της Στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια, του πλαισίου άμυνας για τις των κυβερνοεπιθέσεων που ενεκρίθη από το Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2013 και θα ζητήσω λοιπόν πρώτα από τον κύριο Χέλμπρεχτ να λάβει το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Φωτσίγκα. Θέλω <clears throat> να σας καλωσορίσω και εγώ στη σημερινή συνεδρία. Ελπίζω όλοι να μπορείτε να με ακούσετε. Σήμερα θα ήθελα να σας δώσω μια σύντομη παρουσίαση από την οπτική γωνία της ε, ΕΝΙΣΑ για την οποία η κυβερνοασφάλεια είναι ένα από τα κύρια θέματα αρμοδιοτήτων μας. Ε, οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας είναι η ραχοκοκαλιά της ε, κοινωνίας μας και το βλέπουμε κάθε μέρα όταν χρησιμοποιούμε τάμπλετ, εφή τηλέφωνα, συστήματα τηλεπικοινωνιών, ακόμα και στο σπίτι μας. Αυτό σημαίνει ότι η ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων είναι κεφαλαιώδης για την ασφάλεια όλων των τομέων στην κοινωνία μας. Και φυσικά ξέρετε ότι αν υπάρχουν παραβιάσεις και προβλήματα στις ε, υποδομές της επικοινωνίας μπορούν να προκύψουν σημαντικές απώλειες και ζημίες. Εκατομμυρίων δολάριων πολλές φορές. Θα ήθελα να ξεκινήσω με μια παρουσίαση των τομέων που εμπλέκονται στην κυβερνοασφάλεια. Έχουμε αυτή τη στιγμή ε, κάθε μέρα περιπτώσεις κυβερνο, προβλημάτων κυβερνοασφάλειας. Έχουμε πάρα πολλούς ε, υπολογιστές ε, που χρησιμοποιούμε όλοι μας και εμείς και η κοινωνία των πολιτών. Χρησιμοποιούμε κοινωνικά δίκτυα διαδικτύωσης, το υπολογιστικό νέφος, κάνουμε αγορές στο διαδίκτυο. Αν γυρίσουμε πίσω 15 χρόνια, τότε ξεκίνησε ουσιαστικά να αναπτύσσεται αυτό το είδος υποδομής. Εάν θέλουμε να ταξινομήσουμε όμως όλες αυτές τις ενέργειες κατά της ασφάλειας, πρέπει να μιλήσουμε και για την κυβερνοκατασκοπία, το κυβερνοέγκλημα και την ε, παραβίαση της ασφάλειας. Όταν μιλάμε λοιπόν για τα θέματα της κυβερνοασφάλειας, χρησιμοποιούνται τεχνολογίες και για διαφορετικούς σκοπούς. Είναι πολύ διαφορετική λοιπόν η εικόνα αν δούμε τι συνέβαινε πριν από 15 χρόνια. Γιατί σήμερα με την τεχνολογία που έχουμε μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλαπλούς τομείς η ίδια τεχνολογία για να δημιουργήσει απειλές. Πριν από δύο χρόνια ήταν, έγινε μια κυβερνοεπίθεση σε ένα σταθμό παραγωγής πλουτονίου. Το ίδιο κακόβουλο λογισμικό όπως μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να αντιμετωπίσει όχι μόνο στρατιωτικές εγκαταστάσεις αλλά και πολιτικές εγκαταστάσεις, βιομηχανικές εγκαταστάσεις κτλ. Η πρόκληση λοιπόν που αντιμετωπίζουμε είναι να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη συνεργασία σε όλους αυτούς τους χώρους, ιδίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να σας δώσω λοιπόν ορισμένα παραδείγματα όπου η εμπειρογνωμοσύνη της ΕΝΙΣΑ μπορεί να συμβάλλει σε μεγαλύτερη ασφάλεια. Κάθε χρόνο ε, παρουσιάζουμε μια έκθεση η οποία παρουσιάζει τις απειλές οι οποίες υπάρχουν, τις διάφορες τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, τους τρόπους επιθέσεων και τους στόχους αυτών των επιθέσεων. Για παράδειγμα, άμα έχετε μια ιστοσελίδα, γενικά έχετε εμπιστοσύνη σε αυτήν την ιστοσελίδα. Αν δείτε μια διαφήμιση σε αυτή την ε, ιστοσελίδα, μπορείτε να κάνετε κλικ σε αυτή τη διαφήμιση. Πώς ξέρετε όμως ότι αυτή η διαφήμιση δεν θα σας στείλει σε μια κακόβουλη ιστοσελίδα από όπου θα κατεβάσετε κάποιο λογισμικό το οποίο στη συνέχεια θα επιτεθεί κατά της ασφάλειες του υπολογιστή σας. Ένα άλλο θέμα είναι οι λεγόμενες SERP, οι ομάδες άμεσης απάντησης σε επιθέσεις. Ποιος θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσει μια κατάσταση ανάγκης επίθεσης εάν λάβει χώρα. Τα τελευταία χρόνια Έχουμε δημιουργήσει μια τέτοια ομάδα σε όλες τις ε, πρωτεύουσες της Ευρώπης. Έχουμε βελτιώσει λοιπόν τη λειτουργία τους και έχουμε ένα καλό δίκτυο για ανταλλαγή πληροφοριών σε σχέση με τις απειλές και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις απειλές. Εάν δείτε επίσης και τις διάφορες ασκήσεις που έχουν γίνει και τα γνωρίζετε αυτά τις κυβερνό ασκήσεις που γίνονται ως Επιτροπή Άμυνας και Ασφάλειας. Το 2010 ξεκινήσαμε με τις πρώτες αυτές ασκήσεις επιχάρτου στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Και τώρα οι πανευρωπαϊκές αυτές ασκήσεις κυβερνοασφάλειας είναι μεγάλα, μεγάλες διοργανώσεις. Εξετάσουμε διάφορα σενάρια για το πώς θα μπορούσε να υπάρξει μια παρακόλληση των, της λειτουργίας των υποδομών και θα μπορούσε αυτό να έχει επιπτώσει στην καθημερινή μας ζωή, στη ζωή των επιχειρήσεων και έχουμε διαμορφώσει διάφορες διαδικασίες για αντιμετώπιση περιπτώσεων εκτακτού ανάγκης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κάτι το οποίο επίσης θέλω να σας αναφέρω είναι ότι η εμπειρία μας έχει καταδείξει ότι γινόμαστε όλο και καλύτεροι στο τεχνικό επίπεδο. Αντιμετωπίζουμε τον τομέα τηλεπικοινωνίας ε, για, χρηματο, για τα χρηματοπιστωτικά που και αυτοί ενδιαφέρονται για τα θέματα αυτά το τομέα ενέργειας, τηλεπικοινωνιών. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα αντίδραση σε πολλούς τομείς. Αυτό το οποίο δεν υπάρχει ακόμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι λεγόμενη έδωσα πολέμου. Αν συμβεί κάτι το οποίο πραγματικά είναι μεγάλης κλίμακος, και θυμόμαστε όλοι αυτά που έγιναν στην Εστονία το 2007, είναι απαραίτητο να έχουμε τη δυνατότητα να συντονίσουμε τις ενέργειές μας, να ξέρουμε ποιον θα ξυπνήσουμε στη μέση της νύχτας για να συντονίσει όλες τις ενέργειες. Ποιος επίτροπος, ποιος εθνικός υπεύθυνος θα τα κάνει όλα αυτά. Έχουμε λοιπόν πολύ δρόμο να διατρέξουμε και αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο συζητείται η οδηγία για την ασφάλεια των δικτύων. Θα ακολουθήσει και ένας τριγωνικός διάλογος. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα, εγκριθούν, θα εγκριθεί αυτό το νομοθέτημα. Αλλά το θέμα της διακυβέρνησης των απαραίτητων δομών είναι μια από τις μεγάλες προκλήσεις στην Ευρώπη. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο για τις κρίσιμες υποδομές η Κομισιόν έχει ξεκινήσει με, το, με μια ανακοίνωση το 2009 και έχει αναφέρει πολλά θέματα όπου μπορεί να εμπλακεί η εμπειρογνωμοσύνη της ΕΝΙΣΑ. Έχουμε τώρα την οδηγία για την ασφάλεια των τηλεπικοινωνιών με το άρθρο 8 που αναφέρει την αναφορά συμβάντων. Αυτό αφορά την, ε, τον τομέα των τηλεπικοινωνιών, όταν παραγωγός χάρη μπορεί να υπάρξει ένα κακόβουλο λογισμικό αν πέσουν τα τροφοδοτικά στους ε, διακομιστές κτλ. Αυτά λοιπόν είναι γεγονότα τα οποία τα παρακολουθούμε από πολύ κοντά. Ένα άλλο θέμα είναι το θέμα της κρυπτογράφησης. Αν δείτε τις σημερινές προκλήσεις, υπάρχουν δύο τρόποι να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, τις επιχειρήσεις μας, τις κυβερνήσεις μας. Καταρχήν είναι η ηλεκτρονική ταυτοποίηση και το δεύτερο είναι η κωδικοποίηση. Αν δείτε την πραγματικότητα, εξακολουθούμε να χρησιμοποιούμε τα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία σαν να στέλνουμε προς άλλο ένα στον άλλο. Δεν λαμβάνουμε υπόψη μας το πόσο εύκολα μπορεί να υπάρξει παρεμβολή κάποιου ή πώς μπορεί να παραποιηθεί η ηλεκτρονική επικοινωνία. Με τα ηλεκτρονικά λοιπόν αυτά εργαλεία μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη ασφάλεια και να βελτιώσουμε τη σημερινή κατάσταση. Το τελευταίο στοιχείο που θέλω να αναφέρω είναι τα θέματα της ε, ασφάλειας στην Ευρώπη με τις αποκαλύψεις του Σνόουντεν έγινε φανερό ότι δεν έχουμε τόση ασφάλεια όσο θα μπορούσαμε να φανταστούμε στην Ευρώπη. Υπάρχουν πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά δεν υπάρχουν μεγάλες εταιρείε του μεγεθούς που βρίσκουμε στις ΗΠΑ και στην Κίνα. Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε τις τεχνολογίες ασφάλειας και στον τομέα της πληροφορικής στην Ευρώπη. Αν μπορώ λοιπόν να συνοψίσω όλα αυτά που είπαμε, υπάρχουν διάφορες πτυχές στην αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων και την κυβερνοασφάλεια. Γενικά χρησιμοποιείται σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η ίδια τεχνολογία και γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο τι, ποιος είναι αυτός ο οποίος κάνει τι. Χρειαζόμαστε ε, μια ικανότητα για την ανείχνευση αυτών των επιθέσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν κάποιοι εμπειρογνώμονες για το θέμα αυτό που βρίσκονται και αριστερά μου. Θα πρέπει όμως να προχωρήσουμε σε μια διευρωπαϊκή συνεργασία για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις απειλές και να είμαστε πιο ασφαλείς στην Ευρώπη. Καθηγητά, σας ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Θα επανέλθω σε αυτό το οποίο μας εξηγήσατε αφού μιλήσουν και τρεις ε, εισηγητές. Συζητήσουμε αργότερα. Οπότε επίσης θα έχουμε και την ευκαιρία να θέσουμε κάποιες ερωτήσεις. Και τώρα ήρθε η ώρα για τον κύριο Ρόε. Λάβει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Έχουμε αυτή την ε, παρουσίαση PowerPoint εδώ στην οθόνη πίσω μου, οπότε και θέλω να διαρθρώσω έτσι την ε, ομιλία μου με αυτές τις διαφάνειες. Θέλω να σας ε, μιλήσω για την κυβερνοάμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σχετική πολιτική. Ο συνάδελφος Χέλμπερτ ήδη σας εξήγησε ξεκάθαρα πώς είναι η κατάσταση και εξήγησε το πώς ο ψηφιακός κόσμος ωφελεί αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί και προβλήματα. Και έχουμε όλο ένα και περισσότερα περιστατικά που εκμεταλλεύονται το ψηφιακό κόσμο και οι εγκληματίες. Την επόμενη διαφάνεια μπορεί να δει κάποιες πληροφορίες όσον αφορά το παγκόσμιο πλαίσιο. Το, ο, ο κυβερνοχώρος θεωρείται ο πέμπτος χώρος ε, σε σχέση με το που γίνονται οι συγκρούσεις, οι αναμετρήσεις, οι πόλεμοι. Έχουμε επίσης και τις ε, αποστολές της ε, ΚΕΠΑ Οπότε, γι' αυτό και θα πρέπει και να υποστηριχτούν οι δομές της ΚΕΠΑ. Για να πάμε τώρα στην επόμενη διαφάνεια. Εδώ μπορείτε να δείτε ποια είναι η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλα αυτά. Ίσως θυμάστε ότι τον Φεβρουάριο του 2013 είχαμε την πρώτη στρατηγική κυβερνοασφάλειας. Την είχαν εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο πρώτος εκπρόσωπος εξωτερικής πολιτικής. μπορεί να δείτε εδώ επίσης τους τέσσερις τομείς που καλύπτονται από αυτή την στρατηγική κυβερνοασφαλείας. Το βασικότερο εδώ είναι ότι όλες οι υποενότητες τα διάφορα θέματα τα οποία καλύπτονται από την κυβερνοασφάλεια ασφάλεια καλύπτονται εδώ. Τώρα, για να δούμε ποιοι είναι οι στόχοι της κυβερνόμενας. Σε αυτή τη στρατηγική έχουμε δύο στόχους. Πρώτα-πρώτα να αυξηθεί η αντοχή των συστημάτων μας σε επιχειρήσεις, σε αποστολές, είτε στη έδρα των θεσμικών οργάνων. Στρατηγείο το για να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε τις δυνατότητές μας τόσο να μπορούμε να αντιδράσουμε και να μπορούμε επίσης να αντιμετωπίσουμε τις κυβερνοαπειλές. Τώρα, στην επόμενη διαφάνεια μπορείτε να δείτε κάποια συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2012 2013. Αυτό έγινε όταν ε, ζητήθηκε να επεξεργαστούν μια πολιτική πλαίσιο για την κυβερνοασφάλεια. Όπως ήδη προαναφέρθηκε, όλα αυτά δεν ξεκίνησαν εκ του μηδενός. Ήδη είχαμε και έχουμε κάποια καλά παραδείγματα επιτευγμάτων σε αυτόν τον τομέα που, που ήταν σαν αφετηρία πρώτα-πρώτα η εκπαίδευση συναδέλφων για την κυβερνοασφάλεια ή επίσης ε, το πώς βοηθά η κυβερνοασφάλεια στις θεωρητικές επιχειρήσεις και τη συνεργασία μεταξύ του Φορέα Ασφάλειας EDA και του ΝΑΤΟ για την κυβερνοάμυνα ε, στο κέντρο αριστείας του Ταλίν και άλλα παραδείγματα που είμαι σίγουρος ότι θα τα γνωρίζετε. Θα δούμε τώρα την επόμενη διαφάνεια. Τη, το, την πολιτική πλαίσιο την κυβερνοάμυνα, τον μπορείτε να δείτε τους πέντε τομείς που καλύπτονται. Οπότε θα ήθελα να σταθώ λίγο περισσότερο στις λεπτομέρειες, στην επόμενη διαφάνεια. Πρώτα πρώτα. Το πώς θα αναπτύξουμε τις δυνατότητες των κρατών μελών για την κυβερνοάμυνα. ούτως ώστε να βοηθηθούν οι επικοινωνίες και το δίκτυο πληροφοριών της και πάω όσον αφορά το πόσο λειτουργικά θα είναι. Και έτσι έχουμε αυτό το πρόγραμμα ανάπτυξης των δυνατοτήτων μας ε, και αυτό αφορά τον προγραμματισμό των ε, όσων απαιτείται από πολλά κυβερνάμενος του Προκατημέλη για να συμμετάσχουν σε αυτές τις επιχειρήσεις της θέλουμε να βοηθήσουμε και την ανάπτυξη των δυνατών της ε, επιπλήσης άμυνας για τα project pooling και sharing. Επίσης, συνεργασία μεταξύ των στρατιωτικών cert δηλαδή των τρόπων αντίδρασης. Και επίσης, με αυτό το πλαίσιο πολιτικής θέλουμε να δούμε τι θα γίνει με το δίκτυο επικοινωνιών που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε εδώ μπορεί να δείτε κάποια παραδείγματα. Αυτό το υπαριθμόν 2. Για να δούμε πώς μπορεί αυτές οι δυνατότητες να αφορούν την κάλυψη και τις υπηρεσίες χρηματικής ασφάλειας όσον αφορά την πληροφορική. Και να μπορούμε επίσης να έχουμε και εκτίμηση των κινδύνων. Στην επόμενη διαφάνεια, κάτι άλλο σημαντικό. Επίσης έχει αναφερθεί σε διάφορες εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και αυτό αφορά την συνεργασία στο εφητικό πολιτικού τομέα. Να υπάρχουν δυνατότητες ε, κοινής κυβερνοασφάλειας, δυνατότητες ανταλλαγής των ε, αρίστων πρακτικών. Επίσης θέλουμε εδώ να πετύχουμε μια ευθυγράμμιση όσον αφορά κάποια προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης όπως το Horizon 2020 δύναμη των κανόνων που ισχύουν και επίσης να δούμε πώς η κυβερνοσφάλεια θα ενταχθεί στα προγράμματα τα οποία έχουν διπλή χρήση. Όπως το πρόγραμμα για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό που έχει αυτή την διάσταση λοιπόν της ε, άμυνας και προστασίας. Τέταρτος τομέας είναι το πώς θα βελτιώσουμε την κατάρτιση και εκπαίδευση καθώς και τις ευκαιρίες ε, εξάσκησης. Βλέπετε εδώ κάποια παραδείγματα. Στη δε επόμενη διαφάνεια βλέπετε τον τομέα της εξάσκησης. Να δούμε λίγο πιο κάτω. Βλέπετε εδώ πέρα ένα πρακτικό παράδειγμα του τι μπορεί να γίνει, γιατί ίσως έχετε υπόψη σας κάποια σενάρια τα οποία αναφέρθηκαν από το ε, όπως το Milex και το Multi-Layer. Αυτά τα σενάρια εξάσκησης. Και εδώ έχουμε κάποια συγκεκριμένα πρακτικά ζητήματα, δηλαδή το πώς θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι προετοιμασμένη για κάποια πιθανή επίθεση ή απειλή. Η επόμενη διαφάνεια αφορά την διεθνή συνεργασία. Εδώ έχουμε το ζήτημα της συνεργασίας με το ΝΑΤΟ. Αλλά και με τον ΩΣΑ. Τον ΟΑΣΕ, συγγνώμη. Οπότε βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπάρχει αυτό το ζήτημα το οποίο καλύπτουμε, το οποίο έχει ανακύψει σε διάφορες εκθέσεις πάλι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να, για παράδειγμα, θυμάμαι το ψήφισμα, την έκθεση του κ. Κέλλαμ το 2010, όπου θίγει αυτό το ζήτημα. Στην επόμενη διαφάνεια τώρα. Εδώ αναφέρομαι στο πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ήδη είπαμε ότι αυτό το πλαίσιο πολιτικής ε, αποφασίστηκε τον Νοέμβριο, αλλά εμείς επίσης θέλουμε να κάνουμε και μια έκθεση πρόοδου. Ιούνιο και Ιούλιο ένα τότος έτους. Θα την παρουσιάσουμε τότε και οπότε εδώ και θα καλύψουν το θέμα της ε, κυβέρνου άμυνα στην από τα ζητήματα, τα οποία επίσης πρόκειται να καλυφθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αυτό το οποίο θα λάβει χώρα τον Ιούνιο φέτος. Εν κατακλείδη, θέλω να σας πω ότι όλα αυτά τα οποία σας παρουσίασα θα πρέπει να τα δείτε με τρόπο εγκάρσιο ή οριζόντιο σε σχέση με ε, αυτούς τους πέντε επιμέρους τομείς που παρουσίασα. Επίσης αυτό το πλαίσιο πολιτικής για την κυβερνάμενη είναι κάτι το νέο. Τώρα θα πρέπει να δούμε πώς θα γίνει η εφαρμογή αυτού. Οπότε έτσι θα, με αυτή τη βάση θα πρέπει να ενεργήσουμε, να δούμε τι θα κάνουμε. Αυτή ήταν η παρουσίασή μας. Σας ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ κύριε Ρόι και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Πίτσερ Ράουντ, διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Άμυνας. Έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε να σας μιλήσω για το θέμα αυτό το τόσο σημαντικό για την ενίσχυση της κυβερνοσφάλειας. Από την απόφαση το 2011 να μπει το θέμα της κυβερνοασφάλειας στο πρόγραμμα της υπηρεσίας μας, έχουν ξεκινήσει πολλές δραστηριότητες και πολλά προγράμματα ιδιαίτερα με το πρόγραμμα ανάπτυξης δυναμικού του 2011 και έχουμε υποστηρίξει μια σειρά από ε, πολιτικές στις οποίες ε, έχει θέσει η κυβερνό ασφάλεια σε σχέση με την ε, ΚΕΠΑ. Πριν περάσω στα θέματα πολιτικής, θέλω να σας δώσω μια επισκόπηση της δουλειάς που έχει κάνει μέχρι τώρα η υπηρεσία μας. Όλες οι κυβερνόδραστηριότητες της υπηρεσίας κινούνται από το από την ομάδα κυβερνοασφάλειας. Πρόκειται για εμπειρογνώμονες από 24 κράτη-μέλη και εκπροσώπους από αντίστοιχα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνέρχονται τρεις φορές το χρόνο για δύο μέρες με στόχο να δώσουν καθοδήγηση για δραστηριότητες και νέους τομείς δραστηριοποίησης. Αποτελεί επίση αυτή η ομάδα μια εξαιρετική πλατφόρμα Ανταλλαγή βέλτιστων των εθνικών πρακτικών στον χώρο της άμυνας. Τα τελευταία τρία χρόνια είχαμε τη δυνατότητα να ολοκληρώσουμε 10 προγράμματα κυβερνοασφάλειας με 2 εκατομμύρια ευρώ ε, δημοσιονομικό όγκο από το λειτουργικό προϋπολογισμό της ε, υπηρεσίας μας. Δηλαδή αφιερώσαμε 10% των ετήσων λειτουργικών μας ε, δαπανών στις δραστηριότητες σχετικές με την κυβερνοάμυνα. Από αυτές δίνω παραδείγματα την καταγραφή των υφισταμένων ε, αντιλήψεων και δυνατοτήτων που υπάρχουν στα κράτη-μέλη για την υποστήριξη της κυβερνοασφάλειας, τη θέσπιση μιας έρευνας κυβερνοασφάλειας, κυβερνοάμυνας καλύτερα, επίσης ανάλυση των αναγκών σε κατάρτιση για την κυβερνοάμυνα της ΚΕΠΑ και πιλωτικά νέα μαθήματα όπου εντοπίστηκαν ελλείψεις, ιδιαίτερα όσον αφορά τα ε, ε, ανώτατα στελέχη της στρατιωτικών δυνάμεων και αρμόδιος για τη λήψη των αποφάσεων, αξιολόγησε της ε, αποτελεσματικότητας της θέσπισης μιας κυβερνού, ενός κέντρου κυβερνού και θα επανέλθω αργότερα. Και έτσι εδώ έχουμε τις βάσεις για μια πιο ανθεκτική λειτουργία και πάμε με την κυβερνοάμυνα, πιο λειτουργική επίσης, που δίνει, σαν παράδειγμα, τρία ε, ε, σεμινάρια κυβερνοάμυνας και ευαισθητοποίηση στην κυβερνοάμυνα για το προσωπικό που οργανώθηκαν στο, στη Λάρισα σε συνεργασία με το κέντρο του Ταλίν με το οποίο είχαμε συμφωνία συνεργασίας από το Μάρτιο του 2013. Έχουμε επίσης ξεκινήσει δύο προγράμματα αξιοποίηση κοινών πόρων, όπως κατάρτιση και ε, δοκιμές και ευαισθητοποίηση σε σχέση με καταστάσεις που έχουν να κάνουν με την κυβερνοάμυνα, με τέσσερα κράτη-μέλη. Πρόκειται για προγράμματα που ξεκινούν σε μια προπαρασκευαστική φάση το 2015 και αναμένεται να το 2000, να φάσουμε μάλλον στη φάση της υλοποίησης το 2016. Έχουμε μετά το 2011 ένα νέο σχέδιο του 2014 για την ε, ανάπτυξη δυναμικού με ιδιαίτερη έμφαση την υποστήριξη των κρατών μελών σε ένα, στην ανάπτυξη ενός ικανού εργατικού δυναμικού κυβερνού με τη δυνατότητα για προληπτική δράση αλλά και αντίδραση σε ζητήματα κυβερνού Έχουμε τα κέντρα, κέντρα βάρους όπως ονομάζονται που έχουν ορίσει τα κράτη-μέλη με στόχο τον καλύτερο συντονισμό του, της κατάρτισης και των ε, εξασκήσεων για την κυβερνοάμυνα με την υποστήριξη των κρατών μελών και όλων των εμπλεκόμενων φορέων, νέα προγράμματα σπουδών και την βελτίωση της δυνατότητας εντοπισμού και καταπολέμησης των ΠΕΑ. Θα ήταν σκόπιμο επίση να αναγνωρίσουμε, να σημειώσουμε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε μόνο με ένα κομμάτι της δουλειάς που χρειάζεται για να αντιμετωπιστούν ε, τα καθήκοντα αυτά και ένα μέρος μόνο των που χρειαστούν. Θα ήθελα τώρα να έρθω στο, στην αξιολόγηση αποτελεσματικότητας. Όπως είπαμε είχαμε το σχέδιο ανάπτυξης δυνατοτήτων του 2011 και μια πρόταση για αξιολόγηση και αξιολόγηση για εννιά επιλογές κυβερνοάμυνας οι οποίες είχαν να κάνουν με το, με το κατώτατο στάδιο του να μην αντιδράσουν καθόλου μέχρι την εγκαθίδρυση ενός νέου και πλήρως λειτουργούντος σε όρους ε, τόσο υλικούς όσο και λειτουργικούς κέντρου κυβερνάς άμυνας για να υποστηρίζονται οι δραστηριότητες της ΚΕΠΑ απευθείας. Με ε, την αξιολόγηση λοιπόν που έγινε εξετάστηκαν οι πόροι, η νομική βάση, το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση που θα απαιτούνταν και η δυνατότητα βιωσιμότητας ενός τέτοιου έργου. Αυτή τη στιγμή η ομάδα σχεδίου, σχεδιασμού της κυβερνοάμυνας εξετάζει την τεχνική αξιολόγηση και δεν δίνει συγκεκριμένη προτίμηση ή σύσταση μιας επιλογής, καθώς αυτό θα ήταν μια επιλογή σε πολιτικό επίπεδο, αλλά αναμένεται να ληφθεί μια απόφαση κάπου στα τέλη του εξαμήνου, ώστε να υποβληθούν οι εκτιμήσεις με την έκθεση στην, ε, στους αρμόδιους για τη λήψη αποφάσεων σε πολιτικό επίπεδο. Η υπηρεσία μας συνεργάζεται στενά με κάθε φορέα αρμόδιο για και εμπλεκόμενο σε θέματα κυβερνοάμυνας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, Κράτη-Μέλη, Συμβούλιο και ούτω καθεξής. Έχουμε ήδη προσφέρει αποτελέσματα στον χώρο της άμυνας στην κυβερνό ασφάλεια, στρατηγική ασφάλεια 2012-2013. Έχουμε, νομίζω, με το πλαίσιο πολιτικής κυβερνοάμυνας μπορέσει να καταγράψουμε το ρόλο που διαδραματίζει η υπηρεσία μας και χωρίς να είμαστε εμείς στο τιμόνι της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας μπορούμε να αποδείξουμε σημαντικό έργο και συνεισφορά. Έχουμε 43 συγκεκριμένες δράσεις καταγράψει με περιορισμένους πόρους υλοποιήθηκαν και είχαν πολύ καλά αποτελέσματα. Μπορέσαμε να ε, προσλάβουμε έναν δεύτερο project officer για πλήρη απασχόληση στην, στην τεχνολογία κυβερνοάμυνας και έχουμε περιορισμένους ακόμη ανθρώπινους πόρους αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ορίσουμε προτεραιότητες. Ε, ο τομέας της ε, πολιτικής με τη στρατιωτική συνεργασία και το εισδητής χρήσεως είναι ίσως ο πιο ελκυστικός, γιατί μπορούμε να μοιραστούμε και ανθρώπινους πόρους και διαδικασίες και το καθεξής. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε τουλάχιστον εκεί που είναι πιο έτοιμες οι διαδικασίες να τις αξιοποιήσουμε και να προσπαθήσουμε από τον Ιούνιο και με τις αποφάσεις του Συμβουλίου να ενισχύσουμε και να εμπλουτίσουμε τη δουλειά που ήδη έχει γίνει. Για να ολοκληρώσω λοιπόν, η υπηρεσία μας ε, κάνει μια δουλειά που στόχο έχει να στηρίξει τους στρατιώτες μας όπου δραστηριοποιούνται, αλλά ταυτόχρονα θέλουμε και να ενημερώνουμε τους αρμόδιους για τη λήψη αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα δουλειά σαν στόχο και ε, ένα από αυτά είναι το σεμινάριο ευαισθητοποίησης για τα θέματα της U4RCI στη Λάρισα. Ε, παραμένει η άμυνα μία από τις κύριες προτεραιότητές μας ε, με τα συμπεράσματα του Δεκεμβρίου και του πλαισίου για την πολιτική άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ κύριε Ράουντ. Ξεκινάμε τώρα τη συζήτηση και ο κύριος Κέλλα με έχει ζητήσει να λάβει το λόγο και πιστεύω ότι θα απαντήσετε ήδη <clears throat> στα ερωτήματα του κύριου Κέλλεν και έτσι και τα δικά μου. Ευχαριστώ πολύ, λέει στα πολωνικά ο κύριος Κέλλαμ. <clears throat> Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τόσο ενδιαφέρουσα αυτή η ενημέρωση σε σχέση με την κατάσταση, την πολύπλοκη κατάσταση της Άμυνα. Σύμφωνα με την απόφαση του Δεκεμβρίου 2013, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Έχει παρουσιαστεί λοιπόν η στρατηγική και περιμένουμε τώρα μέσα στους επόμενους τρεις μήνες να πάρουμε την έκθεση πρόοδου για τα θέματα αυτά. Υπάρχουν κάποια θέματα που εγέρθησαν όταν παρουσιάστηκε η κοινοβουλευτική έκθεση για το θέμα της κυβερνοασφάλειας. Το ένα είναι βέβαια το επίπεδο ετοιμότητος για συνεργασία στα κράτη-μέλη. Η δική μου εντύπωση είναι, σε σχέση με την κυβερνοάμυνα ότι αναρωτιέμαι πόσα κράτη-μέλη έχουν κάποια στρατηγική, κάποιο αμυντικό δόγμα στον τομέα του κυβερνοχώρου. Και αν μπορούμε να είμαστε έτοιμοι να δημιουργήσουμε στρατιωτικές μονάδες κυβερνοάμυνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, υπάρχει πραγματικά μεταξύ των ομάδων ΣΕΡΤ, δηλαδή των ομάδων άμεσης αντίδρασης, υπάρχει κάποια συνεργασία ήδη τώρα. Αναφέρεται ότι φυσικά χαιρετίζουμε τις ε, ενέργειες συντονισμού και συνεργασίας, αλλά υπάρχει κάποια πρόθεση να κάνουμε και κοινέ ασκήσεις με τον ΝΑΤΟ στον τομέα της κυβερνοάμυνας. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα είναι το εξής. Αν η οδηγία για την ασφάλεια των δικτύων εξαιρέσει το δημόσιο τομέα δηλαδή τις ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ δημοσίων υπηρεσιών. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα το οποίο θα μπορούσε να προκύψει σε ό,τι αφορά την ασφάλεια στον τομέα της κυβερνοάμυνας. Ίδιος σε ό,τι αφορά το να καθορίσουμε κοινά πρότυπα στον τομέα της κυβερνοάμυνας και της συνεργασίας στον τομέα αυτό. Ελέγχεται επίσης ότι το 2013 το σχέδιο του Συμβουλίου ήταν να μειωθεί σημαντικά το κυβερνό έγκλημα. Έχει συμβεί όμως κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Άννα Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις σας. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικές, πολύ επίκαιρες για μας. Τα ερωτήματά μου ε, επικαλύπτω λιγάκι με αυτά που είπε ο κύριο Κέλαμα, ο οποίο είναι βέβαια ο πραγματικό εμπειρογνώμων στον τομέα αυτό. Σα έθεσα το ερώτημα για τη συνεργασία μεταξύ των μελών, για το αν υπάρχει ήδη κάποια δημιουργία κέντρων κυβερνοασφάλειας στα κρατημέλη. Το ερώτημα όμως θα προχωρήσω λίγο περισσότερο. Αν λειτουργούν αυτά τα κέντρα, γιατί μπορεί να υπάρχουν στα χαρτιά, δεν ξέρω κατά πόσο είναι λειτουργικά όμως στην πράξη. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά κατά πόσο πιστεύετε ότι υπάρχουν επιπτώσεις από τους δημοσιονομικούς περιορισμούς στα κάτι μελη σε ό,τι αφορά τη δημιουργία αυτών των απαραίτητων εθνικών συστημάτων και κέντρων. Και επίσης, για την ανάγκη να δημιουργήσουμε κέντρα κυβερνοασφάλειας που να υποστηρίζουν τις ε, ενέργειες της ΚΕΠΑ. Και αυτό θα είναι για μένα κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί πολύ προσεκτικά γιατί είναι ένα σοβαρό θέμα. Θα ήθελα να ξέρω κατά πόσο εσείς έχετε ήδη κάνει κάποια σχεδίαση ή κάποια επαναξιολόγηση του τι μπορεί να θεωρηθεί για αυτές τις αποστολές ως κρίσιμη υποδομή. Όχι μόνο στις αποστολές αυτού του είδους, αλλά και μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, στις δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν μπορεί λοιπόν να υπάρξει μια κοινή προσέγγιση στρατηγικού χαρακτήρα για την ε, ε, για τον καθορισμό των ε, κέριων υποδομών σε ό,τι αφορά τις επιθέσεις στον κυβερνόχωρο. Επίσης, <clears throat> σε σχέση με το ερώτημα το οποίο ετέθη για τη χρήση μη επανδρομένων αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται και για εμπορικούς στόχους ακόμα αυτή τη στιγμή. Αν έχει υπάρξει κάποια σκέψη σε σχέση με τις επιπτώσεις που μπορεί να υπάρξουν για τη γενική κυβερνοασφάλεια, αλλά ιδίως για τις αποστολές ε, της σκέπα. Και επίσης, ο κύριος Κέλαμ σας έθεσε το θέμα της σύνδεσης με το ΝΑΤΟ, της κοινή δράσης με το ΝΑΤΟ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτός είναι ο τομέας όπου είχαμε πολλά προβλήματα σε σχέση με τους κύριους εταίρους μας όπως είναι οι Ηνωμένε Πολιτείες. Πώς αυτό επηρεάζει τις ε, ενέργειες που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και το τελευταίο μου ερώτημα. Αντιμετωπίσουμε ένα ε, αναβαθμισμένο επίπεδο απειλών από την τρομοκρατία αυτή τη στιγμή και υπάρχει ανάγκη να ενισχύσουμε και την κυβέρνο ασφάλεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε ποιο βαθμό έχει αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό και κατά πόσο υπάρξη υπήρξε ε, σε ό,τι αφορά την αποκοινού θέση των πληροφοριών που συλλέγουν οι υπηρεσίες πληροφοριών των κρατών μελών που δεν είναι τεχνικά βέβαια από τεχνική άποψη τμήματα των αποστολών της ΚΕΠΑ, αλλά όλο και περισσότερο πρέπει να διαμοιραζόμαστε αυτές τις πληροφορίες για να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη κυβέρνηση ασφάλεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει και η πρόεδρος. Ο Μαρκ Γιούρικ θέλει να λάβει το λόγο ή όχι. Η κυρία κυρια λουζινγκ Ευχαριστώ για την παρουσία σας. συχνά το συζητούμε και το αναφέρατε και εσείς στις ε, παρουσιάσεις σας, ε, το θέμα της άμυνας αποκλειστικά. Να περιμένω δύο λεπτά. Μάλλον καταλαβαίνετε όλοι γερμανικά. Λοιπόν, άμυνα. Η άμυνα βεβαίως σε σχέση με κάποια επίθεση. Θα ήθελα λοιπόν ε, να δούμε τη δική σας την επιθετική στάση ή πώς βλέπετε εσείς την ε, πτυχή της επίθεσης. Υπάρχουν όντως κάποιες ε, αναφορές ότι οι Ηνωμένε Πολιτείες και η Γερμανία μεταξύ άλλων κρατών έχουν αναπτύξει δράσεις επιθετικές ή δυναμικό ανάπτυξης επιθετικών δράσεων και εάν ισχύει αυτό προς ποια κράτη και μάλιστα τις δύσεις ή τι είδους ή σε ποιο βαθμό ε, μπορούμε να πούμε ότι κυβερνοστρατεύματα, παράδοξη χρήση μιας τέτοιας ε, λέξης, αλλά κυβερνοστρατεύματα έχουν ενεργοποιηθεί. Άλλη μια ερώτηση. Θεωρώ ότι έχουμε να κάνουμε μια ανησυχητική στρατιωτικοποίηση του ίντερνετ. Είναι ένα όπλο βέβαια το ίντερνετ και αυτό και μπορεί να αξιοποιηθεί με στρατηγικό σχεδιασμό. Μιλάμε για ΝΑΤΟ, μιλάμε για ασκήσεις, ε, χρησιμοποιείται όλη αυτή η στρατιωτική ορολογία. Διερωτώ με λοιπόν κι εγώ. Πρέπει να δούμε το ίντερνετ και σε όρους εξοπλισμών, μεταξύ άλλων. Σας έχει απασχολήσει ή πρέπει να μας απασχολήσει ενδεχομένως εάν ε, πρέπει να υπάρξει κάποιο είδους ε, σύμβαση ελέγχου των εξοπλισμών στο ίντερνετ. Και τι είδους μορφή θα μπορούσε να πάρει μια τέτοια σύμβαση ελέγχου των εξοπλισμών στο ίντερνετ. Έχω ακούσει κάποιους συμπρογνώμενους να μιλούν για το θέμα αυτό. Γι' αυτό δεν ήθελα και τη δική σας γνώμη και να μας πείτε πώς θα, τι εικόνα θα έδινε αυτή η κατάσταση. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Fronzolica. Ευχαριστώ, λέει η πρόεδρος, με τον κύριο President. Ευχαριστώ, κύριε πρόεδρε. Λες τα πολωνικά. Κυρίες και κύριοι. Μιλούμε για μια στρατηγική κυβερνόμενας ένα πλαίσιο πολιτικής στρατηγικής για την κυβερνάμινα. Ταυτόχρονα όμως μιλούμε για έναν νέο κανονισμό, ε, ο οποίος βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση. Και με αυτόν τον νέο κανονισμό θα αναβαθμίσουμε την υπηρεσία προστασία δικτύων της Ευρωπαϊκής Ένωση. Η εντολή των διαπραγματεύσεων δεν προβλέπει αλλαγή της εντολής της ενίσα της υπηρεσίας προστασίας των δικτύων. Άρα, πώς θα την αναβαθμίσουμε αυτή την υπηρεσία να δεν μπορέσουμε να της δώσουμε περισσότερες αρμοδιότητες, περισσότερες εξουσίες, περισσότερους στόχους και περισσότερα μέσα πολιτικής. Πρέπει να αλλάξουμε την εντολή της, δεν το καταλαβαίνω. Επίσης, κυρίες και κύριοι, πρόσφατα διαπιστώσαμε ότι έχουν υποστεί κάποια ευρωπαϊκά κράτη επιθέσει. Εμεί ω Ευρωπαϊκή Ένωση, βέβαια, ε, ξέρουμε ποιε είναι οι κανόνε εμπλοκή, ξέρουμε ποιοι είναι οι κανόνες ε, του, του, του, πολέμου. Σε κλασικό πόλεμο, όταν κανείς υφίσταται επίθεση, του αντεπιτίθεται, μπορεί κανεί να ε, ε χρησιμοποιήσει και κάποιο αντίπεινα. όλα αυτά όμως στον, κυβερνο, στον κυβερνοπόλεμο πώ γίνονται, γιατί ξέρουμε ότι έχουμε υποστεί επιθέσεις επιθέσει, αλλά δεν κάναμε τίποτα μετά. Ούτε μπορούσαμε να προλάβουμε να, αυτές τις κυβερνοεπιθέσεις και τελικά όλες αυτές οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες από ό,τι φαίνεται δεν είναι πάρα πολύ χρήσιμες για να το θέσω έτσι διπλωματικά και σε ευχαριστώ πολύ. Ε, Εμεί ευχαριστούμε λοιπόν και δίνω το λόγο στον κύριο Γκάλερ. Ευχαριστώ πολύ λέει ο Γκάλερ. Προηγουμένως, στην παρουσίασή σας, αναφέρθηκαν οι ίδιες οι ικανότητες στον τομέα της πληροφορικής. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα κατά πόσο θα μπορούσαμε να έχουμε μια απόλυτα αυτόνομη λειτουργία σε ό,τι αφορά τα δίκτυα υπολογιστών για τις αποστολές της ΚΕΠΑ. Θα μπορούσαμε λοιπόν κάπως αυτό να το εντάξουμε στο πρόγραμμα Horizon 2020. Ε, μέσα στα πλαίσια των προμηθειών που έχουν δημόσιο χαρακτήρα. Ποια είναι η άποψή σας λοιπόν για το αν θα μπορούσαν και τέτοιου είδους ενέργειες να ενταχθούν στο πλαίσιο της προμήθειας δημοσίων ε, αγαθών ή υπηρεσιών. Μήπως η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θα μπορούσε να εξασφαλίσει για τις δικές αποστολές ότι θα έχει το δικό της λογισμικό και υλικό. Ευχαριστώ. Κύριος ε, Ζέμκα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και τους καλεσμένους μας για όλες τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες που μας έδωσαν. Κάτω να έχω δύο ερωτήσεις. Πρώτα πρώτα. Μέχρι τώρα δεν έχουμε απειληθεί από κλασική μορφή πολέμου, αλλά υπάρχουν απειλές στον χώρο Και αυτό το φαινόμενο πιστεύω ότι θα ενταθεί. Γι' αυτό σα ρωτώ πρώτον. Για πέστε μου κύριε Χέλμπρεχτ, μπορείτε να μας ε, πείτε δύο λόγια με περισσότερε λεπτομέρειε όσον αφορά τι δυνατότητε, της ε, υπηρεσία σα, Τι γίνεται από πλευρά ανθρωπίνων πόρων, από πλευρά. Ε, νομικών μέσων κλπ. Πέραν αυτού έχω μια άλλη ερώτηση. Τι σχέδια έχετε και προγραμματίζετε να κάνετε για να εξελίξετε ε, την ε, υπηρεσία σας γιατί όπως ξέρετε υπάρχει πολιτική συγκράτηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Αλλιώ θα πρέπει να γίνει στροφή στα δημοσιονομικά. Όμω τώρα μιλούμε για άμυνα και χρειάζονται επομένω περισσότερη πορεία για την άμυνα. Άλλη μου ερώτηση όσον αφορά την λειτουργία της υπηρεσίας σας, η οποία απαιτεί λειτουργική επιχειρησιακή συνεργασία με τους ομολόγους σας των κρατών μελών. Και σας ερωτώ. Πώς θα υλοποιηθεί αυτή η δέουσα συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Δεν ζητεί άλλο το λόγο, οπότε θα υποβάλω τις δικές μου ερωτήσεις και ίσως έχω μια γύρο ερωτήσεων αφού δοθούν οι απαντήσεις. Ίσως. Προς τον κύριο Χέλμπριχτ έχω μια ερώτηση. Το πρόγραμμα για το διάστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι θα γίνει. Στο αμεσομέρον πρόκειται να υπάρξει κάποιο πλαισίωση αυτού του προγράμματο ούτως ώστε να το προστατεύσουμε από τις επιθέσει και από πιθανή, ε, πιθανό δυναμητισμό. Επίσης, βεβαίως και θα έχετε προσέξει το ότι έχουμε λένε και περισσότερα συμβάντα. λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, λόγω των επιθέσεων των ριζοσπαστών ε, Ισλαμιστών της, ε, του Ισλαμικού κράτους στην Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό, τι σκέπτεστε, τι θα πρέπει να γίνει από τη δική σας πλευρά. τώρα προς τον κύριο Ρόε. Μπορείτε να μας ε, αναφέρετε κάποιους τομείς συνεργασίας με το κέντρο εργασίας του Ιταλίνου. Ε, και αυτό το κέντρο που αναφέρατε επίση που αφορά την κυβερνοασφάλεια. Επίσης, τι σκέφτεστε. Υπάρχει δυνατότητα να εξυγχρονίσουμε το μηχανισμό Αθήνα. όσον αφορά τις αποστολές. Και τώρα για τον κύριο Ράουντ. Μπορείτε να επεκταθείτε λίγο παραπάνω όσον αφορά την ε, συμφωνία μεταξύ, αριστείας μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας ε, Άμυνας. Τι κοινέ δραστηριότητες προβλέπονται. Επίσης, μπορείτε να μας πείτε πώς βλέπετε γενικώ το θέμα των δυνατών των κρατών μελών από πλευράς κυβερνών ασφάλειας. Ακριβώς όπως και ο κ. Ζέμκα, το ίδιο θα ρωτήσω ουσιαστικά, γιατί ξέρω ότι υπήρχε ένα τέτοιο πρόγραμμα με την υπηρεσία, εσωτερικής, ε, με την υπηρεσία Ευρωπαϊκής Άμυνας. Οπότε πώς βλέπετε να ολοκληρώνεται αυτό το πρόγραμμα. Sorry. Έχετε το λόγο. Ας ξεκινήσω για να απαντήσω όσο μπορώ στις ε, ερωτήσεις. Καταρχάς, χαίρομαι ιδιαίτερα για τη συζήτηση. Περνάμε στην πρώτη δήλωση. Όταν γίνεται λόγο σήμερα για διαδικτύο κυβερνοχώρο, όπω όπως όλοι θέλετε να το πείτε, έχουμε να κάνουμε με την άγρια δύση. Ο καθής μπορεί να πράξει ό,τι βούλεται στο διαδίκτυο, χωρίς έλεγχο, χωρίς ρύθμιση. Και διαπιστώνουμε στο καθημερινό μας βίο ότι αν θέλουμε να κάνουμε κάτι αν θέλει κανείς να αποδοθεί σε ένα κυβερνό έγκλημα ή οτιδήποτε άλλο, αν θέλει κανείς να καταπολεμήσει καλύτερα το κυβερνό έγκλημα, δεν μπορεί να βρει άκρη. Και αυτό και ελπίζω να μην κατηγορηθώ για κάποιες δηλώσεις που θα κάνω τώρα, αλλά αυτή είναι η γνώμη μου. Έχει να κάνει με την ε, δομή διαχείρισης του διαδικτύου και ποιος επηρεάζει το διαδικτύο ή τι είδους επίδραση μπορεί να έχει η Ευρώπη από τη δική μας λοιπόν την πτυχή, εμείς εξετάζουμε την κατάσταση από την οπτική της ενίας αγοράς. Προοπτικές, τέσσερα εργασίας, ανάπτυξη κοινωνία των πολιτών και ένα ανοιχτό και ασφαλές διαδίκτυο. Αυτή είναι η δική μας προοπτική. Αλλά όλες αυτές οι εταιρείες, και δεν χρειάζεται να τις αναφέρω, έχουν αναπτύξει ένα επιχειρησιακό μοντέλο τα τελευταία 15-20 χρόνια, έχω ξεκινώντας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την τελευταία δεκαετία όμως έχουν ε, επιταχύνει τους ρυθμούς τους κάποιες κινέζικες εταιρείε και αυτές έχουν καταφέρει να επικρατήσουν στην παγκοσμία αγορά. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό για μας και ξεκινώ από αυτό μια και αναφέρθηκε προς το δυναμικό της πληροφορικής για να λογιστείτε το. στην Ευρώπη έχουμε καλέ τομέα τηλεπικοινωνιών. Είμαστε ισχυροί σε αυτό. Έχουμε καλά έσοδα από τις τηλεπικοινωνίες. Όμως στηριζόμαστε κυρίως σε αμερικανικά και κινέζικα προϊόντα. Εάν οι υποδομές μας για κινητά τηλέφωνα, είτε πρόκειται για το τηλέφωνο, είτε πρόκειται για, την, για το smartphone, είτε πρόκειται για το φορητό υπολογιστή, αν δούμε ότι προέρχονται από τις ΗΠΑ, την Νότια Κορέα, την Ιαπωνία, την Κίνα, συντριπτικά, και αρχίσουμε να μιλάμε μετά για το τι συνέπειες μπορεί να έχει για την άμυνα ή την πολιτική άμυνα, ε, θα έλεγα ότι ο, ως απάντηση ότι ο hacker δεν κάνει καμία διάκριση. ναι για δείτε τι έγινε εκεί. έγινε επίθεση κατά τη Siemens, κατά των μονάδων παραγωγής και η επίθεση μπόρεσε να ολοκληρωθεί μέσω stick USB. Άρα η επίθεση μπορεί να ξεκινήσει εις βάρος πολιτικών δομών, μη στρατιωτικών. Γιατί εκεί δεν έχουμε καμία δυνατότητα. Αν έχουμε να κάνουμε μια παραδοσιακή στρατιωτική επίθεση, διαδικασίες προβλέπονται. Ενώ εδώ ή δεν ξέρουμε ή δεν μπορούμε να διαγνώσουμε από πού προέρχεται η επίθεση, απλώς βλέπουμε να εξελίσσεται κάτι. Παραδείγματα, με βάση ερωτήσεις. Όταν μιλούμε για στρατιωτικές πτυχές ή μη, μη στρατιωτικές δομές, εμείς ασχολούμαστε μόνο με τις κυβερνητικές πολιτικές δράσεις ασκήσεις που αναφέρθηκαν. Ο τομέας της άμυνα αναπτύσσει ασκήσει, όπω και εμείς, μερικές φορές κάνουμε ανταλλαγέ με τους δικού μας, αλλά κάνουμε τις δικές μας ασκήσεις. Κύβερνο έγκλημα που αναφέρθηκε επίση σε μια ερώτηση. Ε, ενισχύεται η παρουσία του. Αλλά λίγα σημαίνει αυτή η πρόταση, γιατί στην ουσία ο εγκληματίας θα πάει εκεί που μπορεί να βγάλει χρήμα. Και δεν χρειάζεται πλέον να σηκώσει όπλο για να ληστέψει τράπεζα. Μπορεί να το κάνει μέσω του ίντερνετ, να βγάλει πιο πολλά λεφτά, με έναν απλό τρόπο που ονομάζεται phishing. Αυτά μπορεί να προσφέρει το κυβερνό έγκλημα. Η Europol μπορεί να σας πιο πολλές απαντήσεις. Για τα μη επανδρομένα αεροπλάνα που αναφέρθηκαν. Σας το είπα και στην αρχή. 8.200 ευρώ κάνει ένα τέτοιο αεροπλάνο, τηλεκατευθυνόμενο, πανεύκολο μπορεί να το αγοράσετε και να το χρησιμοποιήσετε όπως θέλετε. Ποια είναι η διαφορά μέσα στον εκβιασμό, το έγκλημα, στρατιωτική επίθεση. Αν το φορτώσετε και κάτι από κάτω την τρομοκρατία, η ίδια τεχνολογία μπορεί να επιτρέψει σε όποιον θέλει να κάνει το οτιδήποτε. Άμα μπορέσει να σηκώσει το αεροπλάνο στον αέρα αυτό, δεν τον σταματάει κανείς. Για την ε, ανταλλαγή πληροφοριών, Εδώ έχουμε να κάνουμε ένα τομέα που έχει να κάνει με την εθνική ασφάλεια και άρα είναι πιο δύσκολη η ανταλλαγή. Έγινε λόγος επίσης για τον έλεγχο των ε, συμβάσεων εξοπλισμών. Θα το πω, όσο δεν υπάρχουν μηχανισμοί να συζητηθεί κάτι τέτοιο, Ξεχάστε το, δεν υπάρχει τρόπος. Το πρόβλημα είναι ότι οι πολιτικοί όχι εσείς βέβαια, οι υπουργοί, οι επιτροποί κτλ. θα πρέπει να τον αντιληφθούν κάποια στιγμή. Χαίρομαι που η Μάλστρομ, ε, η Κρούς και η Άστον ε, ανέλαβαν μια πρωτοβουλία ε, η οποία όμως δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα. Αναφέρθηκε η διαδικασία ΝΑΕΣ Ο κλάδος που θα ονόμαζα πολιτική προσέγγιση, κυβερνητικές δομές στα κράτη-μέλη, κρίσιμες υποδομές από την οπτική της πολιτικής προστασίας και καλύτερη συνεργασία. Αυτό κάνουμε. Αυτό σημαίνει ανάπτυξη δυναμικού, δηλαδή σε κάθε κράτος, σε κάθε κυβέρνηση υπάρχει μια αρμόδια αρχή που ασχολείται με την κυβερνοασφάλεια. Αστική, πολιτική όμω δομή, όπως των, υπουργών, των Υπουργείων των Εσωτερικών ή των Τηλεπικοινωνιών, που δεν έχουν αμυντικό τομέα. Η δική μας πόρη. Και μη γελάτε στο σχέδιο καθίδρυσης προβλεπόταν, προβλεπόταν λιγότερο από 50 θέσεις που παραμένουν στο επίπεδο στο πλαίσιο 2014-2019 διότι είχε ζητηθεί ένα 5% περικόπη των πόρων για τις υπηρεσίες. Για μας ευτυχώς δεν επευλήθη περικοπή από τα κρατη και την Επιτροπή. Είμαστε ήδη χεροί να πούμε έτσι. Από 400... 500 εκατομμύρια πολίτες έχουμε μόνο 50 υπαλλήλους. Για το άλλο θέμα δεν μπορώ να απαντήσω γιατί δεν εμπληκόμεθα. Για την Ουκρανία, αν μιλάτε για πρωτοβουλίες των χωρών της ΕΝΙΖΑ. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα στο με αυτόν. Στην Ευρώπη αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες με τα κάρτη της γειτονίας, Τουρκία ή προς το βόρα Νορβηγία ή συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες όπου συμμετέχουμε και σε κάποιες διασκέψεις, αλλά όχι στον τομέα που ζητήσατε εσείς. Ευχαριστώ. Κύριε Ρόη, <clears throat> σας ευχαριστώ. κάποιες παρατηρήσεις σε σχέση με την ε, οικονομική κατάσταση. Μπορώ απλώς να επαναλάβω αυτά τα οποία ελέγχθη από τον προηγούμενο ομιλητή μας. Με την περικοπή των ε, δαπανών έχουν ε, υποφέρει πάρα πολύ οι υπηρεσίες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Είναι πολύ δύσκολο να βρει κανείς πόρους στο τωρινό δημοσιονομικό πλαίσιο και είναι και πολύ δύσκολο να βρει κανείς και ανθρώπινους πόρους που είναι κάτι το οποίο χρειάζεται κατεπηγόντως για τα άλλα θέματα να αναζητήσουμε συνέργειες στην έρευνα και στις τεχνολογικές προσπάθειες στον τομέα της στρατιωτικής έρευνας μαζί με την μη στρατιωτική έρευνα και ανάπτυξη. Εδώ το ορίζον 2020 αναφέρεται ιδιαίτερα στο πλαίσιο της κυβερνοάμυνας, αλλά φυσικά θα πρέπει να ακολουθήσουμε τους κανόνες που έχουμε θεσπιστεί. Θα πρέπει να βρούμε ευφύης λύσεις. για να μπορέσει να γίνει αυτό πραγματικότητα. Σε ό,τι αφορά κοινέ ασκήσεις με το ΝΑΤΟ. Αυτό αναφέρθηκε και είναι γεγονός. <clears throat> Υπάρχουν τέτοιου είδους ασκήσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα ήδη σήμερα. Έχουμε παρατηρητές ασκήσεις του ΝΑΤΟ. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη στιγμή που θα έχουμε μία άσκηση κυβερνό άμυνα στα πλαίσια της ΚΕΠΑ, τότε φυσικά θα εμπλέκονται και οι διεθνείς εταίροι μας βάσει της ε, πολιτικής ασκήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει επομένω ότι θα ληφθεί υπόψη και η πολιτική αυτή ε, πτυχή την οποία ανέφερε και η Πρόεδρος που βέβαια είναι πολύ σημαντικό το θέμα της συνεργασίας και εδώ αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από τη μια μέρα στην άλλη είναι ένα πολύ μεγαλύτερο ζήτημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αναφέρεστε επίσης και στη Συμφωνία Σύνδεσης του Ευρωπαϊκού Φορέα Άμυνας με το αντίστοιχο κέντρο του ΝΑΤΟ. Αυτό θα το αφήσω ίσως στο συνάδελφό μου να το αντιμετωπίσει, αλλά θα ήθελα να πω ότι πράγματι και αυτή η πτυχή αναφέρεται στο πλαίσιο κυβέρνο άμυνας και γνωρίζω ότι υπάρχουν κάποια σχέδια τα οποία είναι σε σχεδιασμό και μπορούν να ληφθούν υπόψη. Για το κυβέρνο έγκλημα. Η αύξηση του κυβέρνου εγκλήματος. Η Europol έχει κάνει μια έκθεση για τα θέματα αυτά πρόσφατα και η έκθεση δίνει σαφή στοιχεία και φαίνεται από τα στοιχεία αυτά ότι αυξάνει η εγκληματικότητα στον χώρο. Πρέπει όμως να υπογραμμίσουμε ότι ορισμένες ενέργειες των κρατών μελών και οι ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνουν ό,τι μπορούν για να αντιμετωπίσουν αυτή την <clears throat> κατάσταση. Και αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο εμεί θέλουμε να προωθήσουμε τόσο πολύ τη σύμβαση της Βουδαπέστης για το κυβέρνο έγκλημα. Γιατί αυτό συνδέεται και με την εξωτερική διάσταση. Οι χώρες οι οποίες δεν έχουν την αντίστοιχη νομική βάση μπορούν να πάρουν σαν έμπνευση αυτή τη σύμβαση για να αντιμετωπίσουν με αποτελεσματικό τρόπο το πρόβλημα αυτό της κυβερνοασφάλειας. Και αυτό συνδέεται και με διάφορες ε, ενέργειες δημιουργίας ικανότητας τις οποίες εμείς θέλουμε να φέρουμε σε πέρας για τη σύνδεση με την τρομοκρατία. Και αυτό θα αντιμετωπιστεί. Και αυτό μετά από τα πρόσφατα γεγονότα, ιδίως τα γεγονότα του Σαλιεμπτό, όλα αυτά μας ε, οδήγησαν σε κάποια σαφή συμπεράσματα στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών και στο Συμβούλιο Εσωτερικών και Δικαστικών και φυσικά έχει αντιμετωπιστεί στις συνεδριάσεις των επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο συνδέεται με πολλά από τα προηγούμενα τα οποία αναφέρθηκαν. Η κυρία Φωτίγκα έθεσε ένα ερώτημα. Το θέμα του υβριδικού πολέμου και το πώς μπορεί να αντιμετωπιστούν τέτοιες ενέργειες. Αλλά αυτό δεν είναι καθαρά θέμα ασφάλειας, Το έχουμε όμως στο μυαλό μας. Και τέλος, για το θέμα της νομοθεσίας η οποία διέπει όλα αυτά. Και εδώ θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι σε επίπεδο διεθνούς δικαίου υπάρχουν οι ρήτρες αυτές στο διεθνές δίκαιο που αφορούν και τις κυβερνοεπιθέσεις. Το θέμα είναι όμως, και εδώ είναι δυσκολία, σε λεπτομεριακό επίπεδο τι σημαίνουν όλα αυτά. Αλλά έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδο, συνεχίζονται οι συζητήσεις, παραδείγματος χάρη στα Ηνωμένα Έθνη, με τίτλο «Κώδεξ Δεοντολογίας» πρότυπα συμπεριφοράς. Και εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τονίσει ότι κατά τη δική της άποψη όλοι αυτοί οι κανόνες θα πρέπει να εφαρμοστούν και εμείς υποστηρίζουμε τις διαδικασίες για πρότυπα συμπεριφορά στον τομέα αυτό. Και επίσης υποστηρίζουμε όλες αυτές τις ενέργειες οι οποίες οδηγούν σε οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Και επομένως υποστηρίζουμε τις προσπάθειες που έχουν γίνει στον ΟΑΣΕ, που είναι και αυτός ένας φορέας με τον οποίο συνεργαζόμαστε, Όλα αυτά βέβαια είναι απλώς εν εξελίξη αυτή τη στιγμή. Όλη η πολιτική κυβερνοασφάλειας είναι εν το γενάστε, εν κινήσει, αλλά νομίζω ότι και αυτή η συζήτηση που κάναμε σήμερα, η ανταλλαγή απόψεων, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, μια σημαντική συμβολή που θα μπορέσει να μας βοηθήσει για περαιτέρω πρόοδο. Ευχαριστώ πολύ. απαντήσω κάποιες ερωτήσεις με τη σειρά που έχω σημειώσει και αν κάποιον ε, παρέλειψα παρακαλώ να μου το υποδείξετε πρώτα πρώτα όσον αφορά αυτήν μας την μελέτη, το έργο το οποίο κάναμε τέλο πάντων όσον αφορά την κατανόηση από πλευράς κατών μελών και δεσμεύων οργάνων των Βρυξελών όσον αφορά τις δυνατότητές τους για την κυβερνοάμυνα. Νομίζω, για να κρύψω τώρα μια, διαφορετικές ερωτήσεις, πολλές ερωτήσεις που υπευλήθησαν, είναι το ότι σε ποια θέση, τι κατάσταση βρίσκονται τα κράτη-μέλη και η απάντηση είναι ότι έχουν αμυντικό δόγμα, έχουν κάποιες ε, διαδικασίες που προλαβαίνονται. Ε, βέβαια, είναι άνηση κατάσταση από κράτο σε κράτο, μερικοί δεν έχουν τίποτα και θυμάμαι τι έγινε για τους υπολογιστέ ε, που υπήρχε προστασία δικτύου. Όμως από την άλλη μεριά υπάρχουν κάποια κρατημέλη που έχουν πολύ σημαντικές δυνατότητες. Αυτό μερικά κράτη-μέλη το έχουν δημοσιοποιήσει, μερικά όχι. Τώρα όσον αφορά επιθετικέ δυνατότητες και σε αυτή την περίπτωση τα Υπουργεία μήνε και, ο, διακυβερνήσει οι και ο τύπος επίσημα σε κάποια ακαδημία είπαν ότι έχουν και τέτοιες δυνατότητε επιθετικές. Άλλοι πάλι διάλεξαν να μην το δημοσιοποιήσουν αυτό. Βέβαια το θέμα πλευρά και κυβερνοάμυνα ποιο είναι. Ότι είναι περίπου, να πω, περίπου κάτι σαν το καινούριο μπαρούτι ούτως υπήν, αν μπορούμε να το συγκρίνουμε με τις ε, εξελίξεις ε, πολεμικών δυνατών τελευταία τρεις-τέσσερις αιώνες. Πάλι κάποιοι καθημερινοί δεν θέλουν αυτό να το δημοσιοποιήσουν, επομένω κάποιοι έχουν τέτοιε δυνατότητε, κάποιοι δεν έχουν, επομένω σε αυτή την κούρσα ε, για την κυβερνοάμυνα, μερικοί είναι πιο μπροστά από τους άλλους. Ακριβώς επειδή πρόκειται για καθαρά εθνική αρμοδιότητα. Οπότε στη σχετική μελέτη που κάναμε είδαμε πού υπάρχουν κενά, τι μπορούμε να κάνουμε, μπορούμε να κάνουμε την διαφορά, κάποια προσθεμένη αξία και γι' αυτό τελικά ασχοληθήκαμε με το αμυντικό δόγμα, με την εκπαίδευση και με τον τομέα της κατανόησης του σε ποια θέση βρισκόμαστε και πώς μπορούμε να μοιραστούμε αυτά τα οποία γνωρίζουμε. Οπότε και από πλευρά τη ε, εκπαίδευση υπάρχουν, ε, είναι άνισα τα πράγματα ο υπολογιστή, είναι ας πούμε η πρώτη γραμμή αμήνη. και ασχολήθηκα με κατάρτιση κάποιων ανωτάτων αξιωματικών. Δεν θέλω να είμαι αγενής, αλλά μερικοί από αυτού είχαν δυσκολία να χειριστούν ένα smartphone. Τι να κάνουμε στον πόλεμο που θα πρέπει να λάβουμε κάποιες στρατηγικές αποφάσεις όπου είναι ισχυρό και πάρα πολύ σημαντικό το κύβερνο στοιχείο. Σε σχέση τώρα με το πώς μπορεί να γίνει με τον ιδιωτικό τομέα. Επιτρέψτε να σας πω τι ισχύει και σε σχέση με την συνεργασία με το ΝΑΤΟ και με άλλους φορείς. Ο παραδοτικός πόλεμος αφορά σύνορα, εθνικά σύνορα, ποτάμια και ωκεανούς, θάλασσες, πυκνές ζούγκλες, όλα αυτά τα οποία μπορούν να αποτελέσουν όριο, σύνορο μεταξύ δύο χωρών, δύο δραστηριοτήτων, δύο λαών. Όμως η κυβερνητική δεν γνωρίζει τέτοια, ε, τέτοια σύνορα μεταξύ δύο χωρών, δύο στρατών, μεταξύ των δύο οχθών. Επομένω θα πρέπει να κάνουμε εδώ πέρα ένα γενετικό άλμα. Φυσικά ακόμα έχουμε κάποια σύνορα, είπαμε για τα κρατη είπαμε για τις ε, δυνατότητες στην κυβερνητική, αλλά τα πράγματα βελτιώνουν, τα πράγματα αλλάζουν και όπου μπορούμε συνεργαζόμαστε. με άλλα θεσμικά όργανα για να μπορέσουμε να ανταλλάξουμε πληροφορίε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γιατί νομίζω ότι εδώ πέρα όλο και περισσότερο υπάρχει η αναγνώριση από του εμπλεκομένου ότι η ανταλλαγή πληροφοριών είναι κάτι το καλό. Άρα θα το συνεχίσουμε. Θα παρακολουθήσουμε τι εξελίξει, θα σα ενημερώσουμε και θα έχουμε και κάποιου είδου ε, κοινέ ε, ασκήσει σε κάποιου τομείς. Εκεί που είναι πιο βαθιά, πιο στενή συνεργασία τώρα, όσον αφορά την κρίσιμη υποδομή, τη σημαντική υποδομή. Σε αυτό που έχω να πω ότι ναι, έτσι είναι. Και πολύ πριν την κυβερνητική υπήρχε. Να, ως παράδειγμα, κοιτάξτε, είμαι στεθετικό, οπότε είναι θυμητό να σας ε, λέω αυτές τις παραμείωσεις, δηλαδή πώς μπορούμε να κόψουμε το νερό από μια πόλη. Πρέπει κάποιους, ε, κάποιους αιώνες θα ρίχνα κάποια ζώα νεκρά και σάπια στη, στη, στη δεξαμενή νερό ε, πιο πρόσφατα θα πήγαινα στο υδραγωγείο και θα έφερα ένα βραχικύκλωμα. Σήμερα θα, μπορώ να το κάνω χωρίς να πλησιάσω το υδραγωγείο, τέλος πάντων την, την εταιρεία υδάτων της, ε, της πόλης. Μπορώ να το κάνω από μακριά. Να βλέπετε επομένως το ότι οι σημαντικές υποδομές παραμένουν. Είναι η υγεία, το νερό, το φαγητό. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά πρέπει να δούμε σε συνδυασμό πώς μπορούμε να τα προστατεύσουμε. Προστατεύσουμε, να υπεραμεινθούμε αυτόν. Όσο καλύτερα μπορούμε. Και σας ξαναλέω, πριν από 4 χρόνια, πριν από 400 χρόνια θα είχαμε το, το στρατό να ρίξει νεκρές αγελάδες μέσα στο, στο υδραγωγείο. Ε, θα υπήρχε μια βόμβα στην ε, πριν από ξέρω, 100 χρόνια, πριν 30 χρόνια, τώρα το κάνουμε από μακριά αυτό το να κόψουμε το νερό. Αλλιώ δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο. Τώρα κάτι άλλο για τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, ε, εξαρτώμεθα από το διάστημα απολύτω και, και από το χώρο. Αλλά χρειάζεται χώρο για τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Επομένω εδώ υπάρχει θέμα κυβερνητική. Οπότε εάν θέλουμε να τα ελέγξουμε, εάν θέλουμε να προστατευτούμε από τα αεροσκάφη αυτά, Μπορεί να είναι μικρά. αυτά που παίζουν τα Χριστούγεννα τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Ωραία, παίζουν εκεί και πολεμικά πλάνα είναι αυτά. Όμως θα πρέπει τελικά να υπαχθούν σε κάποιον έλεγχο της κυβερνητικής. Τώρα, για τη σχέση μας με το κέντρο αριστείας του Ταλίν. Όπως σας είπα, είναι κάτι που με αφορά, με ενδιαφέρει και δεν υπάγεται στο ΝΑΤΟ. Απλώς έχει πιστοποιηθεί, έχει εγκριθεί κάποιο τρόπο από το ΝΑΤΟ. Και συνεργαζόμαστε με το κέντρο αυτό. Ανταλλάσσουμε τις άρθρες πρακτικές και τις πληροφορίες. Και όπως προηγουμένως, θα πρέπει να συνεργαζόμαστε. Ακριβώς το ίδιο ισχύει και για το κέντρο του Ταλίνου αν είναι λίγη πληροφοριών, τα πράγματα εκεί είναι υψηλής ποιότητας. Το έχουμε και την πολυ... πολυεθνική εκστρατεία ανάπτυξη δραστηριοτήτων. Πρόκειται για μια διεθνή εκστρατεία για να βελτιωθούν οι δυνατότητες μας αυτές, αφορούν την κυβερνητική και κατά αυτόν τον τρόπο ανταλλάσσουμε εμπειρίες και με χώρες εκτός ΝΑΤΟ και με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και με πολύ μακρινές χώρες. Και αν θέλουμε αν έχουμε μια βαθιά κατανόηση του τι συμβαίνει, θα πρέπει να σκεφτόμαστε με όρους παγκόσμιους όσον αφορά τις κυβερνό απειλές. Γιατί μπορεί επιτιθέμενος να βρίσκεται σε κάποια χώρα που ποτέ μας πέρασε από το μυαλό. Τελικά, βέβαια όλα από τον άνθρωπο και η άμυνα επίσης είναι θέμα ανθρώπου. Μπαγιούν μόνος πολλά. Και ένα από τους τομείς που μας απασχολεί, που σημαντικοί συνάδελφοι, δεν είναι μόνο η εκπαίδευση προσώπων, και όχι μόνο το να μπορούμε να κάνουμε μια αναδρομή, το να έχουμε κάποιο είδου δυνατότητες ούτως ιατροδικαστικέ. και το θέμα δεν είναι μόνο η άμυνα κατά επίθεση. αλλά όπως λέμε δεν, δεν έχει πάντα την ίδια τύχη ο τρομοκράτης. αλλά θα πρέπει να μπορέσουμε να δούμε τις ρίζες των επιθέσεων, να μπορέσουμε να κλείσουμε την πόρτα σε αυτές τις επιθέσεις. Άρα ποιο είναι το μήνυμα, ότι η διεθνής συνεργασία και η διακριτική συνεργασία θα πρέπει να γίνονται όσο γίνεται ευρύτερα σε αυτόν τον τομέα. Εμείς ευχαριστούμε, λέει η Πρόεδρος. Κύριε, σας ευχαριστώ για τις πλήρες και πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις και τις απαντήσεις στις ερωτήσεις των βουλευτών. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση για την κυβερνοασφάλεια στο εγγύς μέλλον, καθώς το θέμα αρχίζει να είναι πολύ σημαντικό και επίγον. Θα χρειαστεί να το συζητούμε τακτικά. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Και αγαπητοί συνάδελφοι, μην φύγετε. Ξεκινάμε μέσω στο επόμενο θέμα. Με την έκθεση Πάσκου. Ladies and gentlemen, please be... Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. Mm. Please take your seats. We start next. Είστε παρακαλώ, θα ξεκινήσουμε με το επόμενο θέμα αμέσως. Πρώτη εξέταση της εκθέσεως του κυρίου Πάσκου. θέμα στρατηγική και στρατιωτική κατάσταση της λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας κατόπιν της προσάρτησης της Χερσονήσου της Κρυμαίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία. Κύριε Πάσκο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Είναι ακριβώς η επέτειος της προσάρτησης πριν από ένα έτος έγινε αυτοί οι προσάρτες και κάποιοι το γιορτάζουν κιόλα. Αν διαβάσετε την σημερινή Washington Post ή την χθεσινή, ο κύριος Πούτιν καφιέται ότι ήταν μια μεγάλη επιτυχία ως μεγάλος στρατιλάτης μπόρεσε να επιτύχει αυτήν την στρατιωτική επιχείρηση προσάρτηση της Κρυμαίας και για πρώτη φορά αποδέχεται ότι αυτά τα άγνωστα άτομα ήταν πράγματι πράκτορες των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων, γιατί εμείς ποτέ δεν μπορούσαμε να φανταστούμε κάτι τέτοιο, ότι θα μπορούσε να γίνει μια τέτοια απόκρυψη από τις ρωσικές αρχές. Αν δείτε λοιπόν τώρα το βόρειο μέτωπο και το νότιο μέτωπο αυτών που συμβαίνουν στην Ανατολική Ευρώπη σήμερα. Βλέπουμε ότι στο βόρειο μέτωπο, εκεί που βρίσκονται οι βαλτικές χώρες, είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε την ε, ανεξαρτησία και την ασφάλεια των χωρών αυτών. Είναι χώρες οι οποίες στο παρελθόν είχαν σταθεί τμήμα της Σοβιετικής Ένωσης και δεν ξέρουμε μέχρι πού θα φτάσει η ρωσική ρεκονκουίστα προσπάθηση ανάκτηση των εδαφών της Σοβιετικής Αυτοκρατορίας. Αν δείτε όμως και στο Νότο, βλέπετε ότι με την παράνομη προσάρτηση της Κρυμαίας υπήρξε μια μεγάλη στρατηγική μεταβολή. Αυτό είναι κάτι το συγκεκριμένο που έλαβε χώρα. Αυτό το έδαφος έχει ενσωματωθεί στη Ρωσική Ομοσπονδία και έχει τώρα το ίδιο νομικό καθεστώς όπως και το Καλίνιγκρατ, η Κενιξφέργη δηλαδή. Και το να ενσωματώσει όλη την ε, Χερσόνησο και όχι μονάχα την Σεβαστούπολη ή κάποιες άλλες βάσεις που είχε χρησιμοποιήσει προηγουμένως ο Ρωσικός στρατός, δίνει τη δυνατότητα να έχει ένα νέο Καλίνιγκρατ στην Μαύρη Θάλασσα η Ρωσία. Έχει λοιπόν τώρα δύο προκεχωρημένα ε, προχωρημένες βάσεις, μία στη Βαλτική και μία στη Μαύρη Θάλασσα. Και καταλαβαίνετε τι σημαίνουν όλα αυτά. Δεν έχει τελειώσει βέβαια αυτή η διαδικασία. Η Ρωσία προσπαθεί με τη συμφωνία Μίνσκ 2 να εξασφαλίσει ότι θα υπάρχει κάποιος διάδρομος που να συνδέει το, το ελεγχόμενο από τη Ρωσία έδαφος της Ουκρανίας και την Κρυμαία και εκεί πέρα είναι κομική σημασία η Μαριούπολη για αυτό το στόχο και επίσης θέλει να δημιουργήσει και ένα άλλο διαβλό από την Κρυμαία στην υπερνηστερία και εκεί το αντίστοιχο της Μαριούπολης είναι η Οδυσσός. Αυτές οι θεωρίες λοιπόν δεν έχουν οδηγήσει και σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, όπως στην περίπτωση Μαριούπολης. Αυτό λοιπόν το οποίο έχει συμβεί μέσα σε ένα χρόνο και μόνο στην Κρυμαία είναι ότι είχαμε κάποιες ε, βάσεις για το ρωσικό στόλο, δύο-τρία αεροδρόμια όπου υπήρχαν αεροπορικές βάσεις για την άμυνα της περιοχής υπήρχαν πύραυλοι εναντίον ε, πλοίων με βραχίβελνικες και υπήρχε μια μικρή αμυντική δύναμη μια κάποια δύναμη πεζοναυτών, μια ταξιαρχία. Στο παρελθόν έτσι ήταν και μέσα σε ένα χρόνο έχουν αλλάξει όλα αυτά. υπάρχει μια αύξηση από 2 με 3 αεροδρόμια υπάρχουν 6 με 9 αεροδρόμια έχουμε δύο ταξιαρχίες αντί για μία και αν λάβει υπόψη κανείς το γεγονός ότι θα πάρει τις φρεγάτες Μιστράλ ενδεχομένως η Ρωσία, η Ρωσία αποκτά μια πολύ σημαντική δύναμη για να μπορεί να κάνει ε, αμφίβιες επιχειρήσεις στην περιοχή. <clears throat> Έχουμε ε, αεροσκάφη τα οποία μπορούν να οπλιστούν με πυράβλους κρούζ, κάτι το οποίο που θα αυξήσουν σημαντικά την ακτίνα δράσης της και με τον τρόπο αυτό μπορεί να φτάσει μέχρι τα όρια της ε, Βουλγαρίας και της Ρουμανίας και από εκεί, αν εκτοξευθούν αυτοί οι πυραυλοί μπορούν να χτυπήσουν και το Στρασβούργο. Και φυσικά μπορούν να επιτεθούν και κατά της Μέσης Ανατολής προς την άλλη κατεύθυνση με αυτή την αεροπορία με τους πυραύλους κρούζ. Η στρατηγική αεροπορική δύναμη βέβαια της Ρωσίας δεν ήταν απαραίτητο να εδράζεται στην Κρυμαία, δεν χρειαζόταν κάτι τέτοιο. Δεν κερδίζει κανείς με μεταφορά της αεροπορίας κατά 100 χιλιόμετρα μεγαλύτερο βεληνικές εναντί της Δύσης. Αλλά ξέρετε ότι σε ό,τι αφορά τον εξυγχρονισμό του στόλου της Μαύρης Θάλασσας και εδώ υπάρχει αυτό το σχέδιο που αναφέρεται εδώ στην έκθεση, 6 νέες φρεγάτες, 6 νέα υποβρύχια και ένα σύστημα άμυνας κατά ε, πολεμικών σκαφών με πύραυλους και το οποίο έχει μεγαλύτερο βεληνικές τώρα και το οποίο μπορεί να καλύψει όλη την μαύρη θάλασσα με τα αμυντικά αυτά πυραυλικά συστήματα που έχουν τη βάση τους στην Κρυμαία. Όλα αυτά τα συστήματα λοιπόν μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε στην ξηρά είτε να επιβιβαστούν σε ένα σκάφος και μπορείτε αμέσως να καταλάβετε πώς διευρύνεται το βελληνικό τους τα τρία τέταρτα του εναέριου χώρου στη Μαύρη Θάλασσα είναι υπορωσικό έλεγχο. Η Τουρκία, η οποία μπορεί να αξισορροπήσει σε επίπεδο ναυτικών δυνάμεων την Τουρκία, δεν έχει τη δυνατότητα να είναι ισόρροπο βάρος με τη Ρωσία σε ό,τι αφορά τα μαχητικά αεροπλάνα. Και νομίζω ότι βλέπετε ότι η στρατιωτική ισορροπία στην περιοχή έχει αλλάξει προς όφελος της Ρωσίας, παρά το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ διατηρεί την γενική του υπεροχή, αλλά με υπόψη και τα άλλα ε, οπλικά συστήματα που μπορούν να κινητοποιηθούν από άλλες πλευρές της Μαύρης Θάλασσας. Το ΝΑΤΟ έχει πάρει μέτρα για να εξασφαλίσει ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια, ασκήσεις εναλλαγής στρατευμάτων, δεν μιλάμε για μεγάλες ε, δυνάμεις. Θα λάβει χώρα τώρα μια άσκηση στη Ρωσία με ε, άρματα μάχης και θωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού που θα συμμετάσχουν σε αυτές τις ε, ασκήσεις. Αυτή είναι η απάντησή μας λοιπόν στα τεκτενόμενα. Αυτό που έχουμε συζητήσει και η κυρία Φωτίκα και άλλοι συνάδελφοι, επίσης και η Άννα ήταν μαζί μας στη Ρήγα συζητήσαμε τα θέματα του υβριδικού πολέμου, που είναι αυτό το οποίο με μεγάλη πτυχία έχει εφαρμόσει η Ρωσία μέχρι το Μάιο του 2014 και στην Ουκρανία αλλά και στην Κρυμαία και πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτή η δυνατότητα υβριδικού πολέμου που κινητοποιεί η Ρωσία. Αν μιλήσουμε για αποκλιμάκωση τώρα, <clears throat> Είναι επιθυμητή η αποκλιμακώση, αλλά όλα εξαρτώνται από το τι θέλει να κάνει η Ρωσία, αν θα εφαρμόσει ή όχι τη συμφωνία του Μίνσκ, αν θα εξακολουθήσει να σπρώχνει στην Ουκρανία ή όχι. Όλα λοιπόν εξαρτώνται απόλυτα <clears throat> από το τι θα γίνει στην Ουκρανία. Και νομίζω ότι κατανοείται ότι αυτό το οποίο είναι τελείως απαραίτητο τώρα είναι ότι ακόμα και αν προκύψει κάποια αποκλιμάκωση, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την στρατηγική εξασφάλιση. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να εμπιστεύεται κανείς τη ρωσική ηγεσία κάτω από αυτές τις ε, συνθήκες. Και έχω λοιπόν ε, όλα αυτά τα στοιχεία στο έγγραφό μου, δεν χρειάζεται να σας τα πω βέβαια, τα ξέρετε πολύ καλά όλα αυτά τα πράγματα, ξέρετε τι λένε οι Ρώσοι, τα απεικονίζω αυτά και στο έγγραφό μου, πώς αντιμετωπίζουν τις επικρίσεις της Δύσης. Ο πόλεμος της προπαγάνδας καλά κρατεί. <clears throat> και εδώ θα πρέπει να το λάβουμε και αυτό υπόψη μας. Αυτά ήθελα λοιπόν να σας πω και είμαι έτοιμος τώρα να ακούσω αυτά που αυτά που θα πούν οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Θα πρέπει να δώσω το λόγο στους και οδησηγητές. Ο κύριος Γκάλερ, εκ μέρους του κύριου Λάντσπεργκης, αν δεν απατώμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ τον Γιάννη Πάσκου για την έκθεση. Ο Γαβρίλος Λαντσπέρκης δεν μπορούσε να έρθει και με παρακάλεσε να σας διαβάσω την ε, δήλωσή του. που λέει ότι συμφωνεί και υποστηρίζει το σχέδιο που παρουσιάζεται. Λέει ότι έχει αλλάξει ριζικά η κατάσταση σχετική με την ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα λόγω της επίθεσης της ε, Ρωσίας στις βάρος της Ουκρανίας καταγράφεται πιστά στο σχέδιο. Η πραγματικότητα αυτή η Ρωσία επέτυχε να αλλοιώσει την ε, εικόνα της ασφάλειας στη Μαύρη Θάλασσα με μια επίθεση απρόκλητη. Για την ε, γεωργία λέει ο κύριος Λαντσβέρκης, υπάρχει ο κίνδυνος και ταυτόχρονα με την προσάρτηση αυτού του μέρους του κομμάτι της Ουκρανίας πρέπει πια να έρθει η ώρα της αφύπνισης. Και πια πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της Ρωσίας, να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας με τον ΝΑΤΟ και τους ιδιωτικούς συμμάχους. Έχουμε στη χέρια μας αποτρεπτικό στοιχείο και πρέπει για τη Ρωσία να καταστεί σαφές ότι πρέπει να υλοποιηθεί πλήρως η συμφωνία του Μίνσκ. Mm. Ιδάλλως θα ενισχυθούν οι κυρώσεις συμπεριλαμβανομένων και νέων κυρώσεων αν δεν επιστρέψουν την Κρυμαία. Αυτό μάλιστα αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα της αντίδρασής μας. Πρέπει όλα τα μέλη να ε, προσυλλοθούν στην υλοποίηση των κυρώσεων για δίποτε συνεργασία στο χώρο της άμυνας με τη Ρωσία. Αποκλείεται μέχρι ότου αποσυρθούν τα στρατεύματά τους από την Ουκρανία, μέχρι ότου πάψουν να προσφέρουν βοήθεια σε τρομοκράτες, μέχρι ότου αποκαταστήσουν επιστρέψουν τον έλεγχο των συνόρων και από την ε, Ουκρανική πλευρά. Ταυτόχρονα για μας δεν υπάρχουν τυπικοί περιορισμοί για την περαιτέρω σωτική συνεργασία με την Ουκρανία. Αυτό πρέπει να δηλωθεί απερίφραστα. Δηλαδή κάθε κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει μόνο του το βαθμό της στρατιωτικής συνεργασίας με την Ουκρανία. Παράλληλα λέει ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την ε, ε, ανθεκτικότητά της και να συνεχίσει το στρατηγικό σχεδιασμό σε σχέση με την ε, Μαύρη Θάλασσα, να ενισχύσει την ΚΕΠΑΣ της ευρωπαϊκές πολιτικές γειτονίες, να, να σχεδιάσει συγκεκριμένα μέτρα και απτές αντιδράσεις σε γεγονότα και σχετικές πληροφορίες που στρέφονται κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εταίρων της που βρέχονται από τη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας. Από την ανάληψη των καθηκόντων από τον Πούτιν έχει μπει σε μία κατάσταση υπερδύναμης. Προσπαθεί να ανακτήσει τον ζωτικό του χώρο η Ρωσία και βλέπουμε αυτό να με μια στρατηγική στις γειτονικέ χώρες αλλά και πέραν αυτών και το ζήτημα δεν είναι μόνο η Ουκρανία αλλά η αντιπαράθεση μεταξύ αυταρχισμού και των αξιών των φιλελεύθερων κρατών που διεκδικούν η ειρηνική σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος μας θα είναι να αντιδράσουμε στην πρόκληση αυτή. Αυτή ήταν η δήλωση του συναδέλφου Λαντσπέρκης. Και σταματώ εδώ. Ευχαριστούμε, κύριε Γκάλερ. Κύριος Γιούρικ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα-πρώτα, να συγχαρούμε τον εισηγητή. Να ευχαριστούμε για αυτό το κείμενο αλλά και για την πρωτοβουλία του γιατί πολλές φορές δεν ξέρουμε ποια είναι τα όρια μεταξύ έρευνας και πολιτικής δράσης. Γιατί θα πρέπει τα κείμενά μας να προκαλούν πολιτικό προβληματισμό. Γι' αυτό σας λέω ότι η έκθεση αυτή είναι πολύ αξιόλογη. Ξεκινώ από το πιο σημαντικό, κάτι το οποίο αναφέρεται στο κείμενο και κατόπιν θα προχωρήσω σε άλλα ζημία. Πρώτα πρώτα. Αυτό το συμπέρασμα ότι η προσάρτηση της Κρυμαίας έχει μεταβάλει ε, το στρατηγικό στάτους quo στην ε, ε, περιοχή. Ναι, αυτό, αυτό το συμπέρασμα έχει δυναμικό χαρακτήρα και επομένω θα πρέπει και εμείς να προβούμε σε αλλαγές στη δική μας πολιτική. Ήταν ε, πολύ σημαντική αλλαγή που έγινε εκεί στο Status Η θεωρήσαμε ότι στη Σεβαστούπολη ήταν προσωρινή διαμονή ο ελιμενισμός τέλο πάντων του Ρωσικού στόλου, κατόπιν έγινε η κατάληψη και η προσάρτηση της Κρυμαίας κλπ. Οπότε τώρα πρέπει να δούμε πώς το ΝΑΤΟ αποφασιστικά θα τοποθετηθεί. για να βοηθήσει τα όμορα κρατημέλη, τα κρατημέλη που συνορεύουν δηλαδή με την ε, Κρυμαία, δηλαδή την Ρουμανία κυρίω. Να διευρυνθεί δηλαδή το πώς μπορούμε να αναλάβουμε κάποιες ε, στρατηγικές ε, πρωτοβουλίες ασφάλειας και άμυνας γιατί νομίζω φυσικά ότι όλα τα κάτι μέλη της Ένωσης είναι και μέλη του ΝΑΤΟ. Βλέπουμε μόνος τι έγινε τώρα στην ε, Κρυμαία από πλευράς ε, ανθρωπιστικής. Υπάρχει πρόβλημα εκεί με τους Τατάρους της Κρυμαίας, θα πρέπει να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις εκεί, αλλά θα πρέπει να βοηθήσουμε και τους Ουκρανούς της Κρυμαίας. να μην γίνουν τα πράγματα ακόμα χειρότερα. Άρα θα πρέπει να δούμε το όλο το οποίο και να μην ξεχνούμε ότι τη σύγκρουση αυτή την χρησιμοποιεί η Ρωσία. Τη χρησιμοποιεί για να ασκήσει πίεση. Να πιέσει διάφορα κράτη. Και όπως ξέρετε ήταν έτοιμη να χρησιμοποιήσει πυρηνικά και θα τα χρησιμοποιούσε κατά χώρα που δεν έχει πυρηνικά. Και αυτό πρέπει να μπει στην έκθεση. Επίση, θα πρέπει να πούμε περισσότερα στην έκθεση για την γεωργία. Γιατί είναι κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία. Και σας υπενθυμίζω το τι κάνει η Ρωσία ούτως ώστε να μονιμοποιήσει εκεί την ε, παρουσία της. Άρα και εμείς θα πρέπει να ρυθμίσουμε την θέση μας ως προς την γεωργία. αν συνεχιστεί η κατάσταση αυτή στην Κρυμαία, τότε θα πρέπει να αναλάβουμε συγκεκριμένα διαβήματα και έτσι να επιταχύνουμε την ε, προσέγγιση, την ένταξη της ε, Γεωργίας στο ΝΑΤΟ. Αυτό θα ήταν ένας έξυπνος τρόπος να πιέσουμε τη Ρωσία. Άλλο, τρίτο. Είναι κάτι που το έθιξε ο κύριος Γκάλερ. το πώς θα βοηθήσουμε με οπλισμό την Ουκρανία. Δεν υπάρχει πια το εμπάργκο για τους εξοπλισμούς. Επομένως, να βοηθήσουμε και αυτή την πλευρά την Ουκρανία. Επίσης, πέραν της στρατηγικής αυτής της βοήθειας, να θα πρέπει και στην, στο κείμενο της έκθεσης μέσα να απευθύνουμε μια έκκληση ούτως υπήν. Έκλεισε προς όλους όσοι θέλουν να πουλήσουν πολεμικά πλοία στην Ρωσία να μην το πράξουν. Επομένως, ανεξαρτήτως του τι θα γίνει τους αμέσως επόμενους μήνες, δεν θα πρέπει να αναλυθούν τέτοιες ενέργειες από τις χώρες που είναι εταίροι μας. Επίσης, θα πρέπει να επανεξετάσουμε τι γίνεται με το Ναμπούκο, τον αγωγό. Γιατί το project αυτό ήταν επιτυχία, από, αποτυχία από πλευράς μας. Γιατί αν αυτό υλοποιείται, τότε θα είχαμε ενεργειακή αυτάρκεια σε χώρες τη ε, κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Επομένω, θα πρέπει να αποτελέσει το, το θέμα αυτό, να αποτελέσει προτεραιότητά μα. Επίση, να πείσω την προσοχή σα ε, στο πρόβλημα των Ουκρανών και Τατάρων τη Κρυμαία. Θα πρέπει να υπάρχει πέρα μια αποστολή από την κοινότητα. Μονίμως να παραμείνει εκεί και να παρακολουθεί το τι γίνεται με του πληθυσμού αυτού στην Κρυμαία. Και να μην ξεχνούμε το τι γίνεται σε τέτοιε συγκρούσει. Πολλέ φορέ αυτέ οι συγκρούσει ε, χρησιμοποιούνται για να αποσταθεροποιεί την κατάσταση στα κατεχόμενα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι έχουμε και μια επόμενη συνεδρία 24 Μαρτίου με εκπροσώπους τατάρων της Κρυμαίας συμπεριλαμβανομένου και του κυρίου Τζέμιλεφ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στο σκιώδη εισηγητή των Πρασίνων, του κύριο Ταράν. Πρόεδρε, ευχαριστώ και πολύ σύντομα. Είναι πολύ σημαντική έκθεση και ο κύριος ε, Πάσκο έχει κάνει καλή δουλειά. Οφείλω να κάνω τη σχολεία μου από την οπτική των πρασίνων. Κάποια άρθρα μας προβληματίζουν και θα θέλαμε πιο συγκεκριμένη διατύπωση για να μπορέσουμε να διατυπώσουμε το σωστό μήνυμα για τους στρατηγικούς εταίρους όπως λέγαμε πριν τώρα στρατηγικούς αντιπάλους. Μη τυχόν και αντιδράσουν υπερβολικά κλιμακώνοντας τη στρατιωτική κατάσταση. Όπως είπε και ο κύριος Κάλλαρ τώρα, η στρατιωτική συνεργασία δεν είναι πια ζήτημα. Στη Ρουσία. Όμως η Γαλλική Δημοκρατία έχει πρόβλημα με δύο πολεμικά σκάφη Μιστράλ. Ίσως ε, θα μπορούσαν να έχουν επανασχεδιαστεί για άλλη χρήση. Ευρωπαϊκή άμυνα, παραδείγματι. Αντί να πάνε εκεί που θα έπρεπε, που είχαν ταχθεί αρχικά. Όταν μιλούμε για κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας, εμείς πράσινοι λέμε ότι δεν ε, περασπιζόμαστε εδαφικά. Δεν κάνουμε εδαφική άμυνα. Και όταν μιλούμε για ΝΑΤΟ, πρέπει να έχουμε υπόψη ότι δεν είμαστε κοινοβουλευτική συνελεύση του ΝΑΤΟ. Δεν μπορούμε να πάρουμε με τόση ευκολία όσο η κοινοβουλευτική συνελεύση του ΝΑΤΟ τέτοιου είδου αποφάσει δηλαδή. Εν τέλει, με προβληματίζει το άρθρο 18 που καλείται η Ουκρανική κυβέρνηση να αξιοποιήσει κάθε μέσον στη διάθεσή της για να διερευνηθούν εγκλήματα πολέμου που έχουν ενδεχομένω διαπραχθεί ε, στην Κρυμαία. Νομίζω ότι είχε αρκετές δυσκολίες η κυβέρνηση της Ουκρανίας στην διερεύνηση εγκλημάτων στην ε, Κρυμαία. Αλλά θα πρέπει να εξηγήσουμε τι σημαίνουν αυτά που γράφουμε. Αυτά είναι ολίγης. Εκφράζω και την... το θαυμασμό μου προς τον εισηγητή που ανέλαβε ένα τέτοιο θέμα. Είχαμε ένα αρκετά μετριοπαθές ψήφισμα την προηγούμενη εβδομάδα για τη δολοφονία του Νέμζοφ. Ο Υπουργός των Εξωτερικών από την ε, Ρωσία αντέδρασε, ονομάσουμε ονομάζοντας μας ιστερικούς. Κάτι τέτοιο πρέπει να περιμένουμε και για το επόμενο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Στούνη και εγώ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ να ευχαριστήσω τον συνάδελφό μας ε, τον Ιώαν Πάσκου για τη θαυμάσια αυτή και ιδιαίτερα επίκαιρη έκθεση. Για όλους μας νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να καταλάβουμε τι σημαίνει η προσάρτηση της Κρυμαίας σε όλους μας και όχι μονάχα, όχι για την Ουκρανία και για τις όλες χώρες που είναι όμορες της Μαύρης Θάλασσας. Δεν είναι μονάχα μια πολιτική αλλαγή δεν είναι προφανώς μονάχα μια παράνομη πράξη που δεν θα αναγνωρίσουμε. Η πραγματική αλλαγή αφορά την πρακτική μας κατάσταση ασφάλειας και αυτό εμπλέκει όλους μας. Όπως είπατε, η Κρυμαία έχει γίνει βάση για περαιτέρω ρωσική επέκταση. Δεν είναι μονάχα πιθανό, είναι πολύ πιθανό και αν λάβουμε υπόψη ότι για πάρα πολύ καιρό έχουμε αγνοήσει την ε, ενίσχυση του ρωσικού στόλου και των στρατιωτικών δυνάμεων της Ρωσίας στην Κρυμαία και τη Μαύρη Θάλασσα, αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι να φέρουμε και πάλι στο προσκήνιο της προσοχής μας το θέμα αυτό. Ο κύριος Τάραντα ανέφερε το εκρεμές θέμα των φρεγατών Μιστράλ. Η γαλλική κυβέρνηση δεν είπε ότι δεν θα παραδώσει αυτά τα πλοία. Η απόφαση αυτή θα είναι κομβικού χαρακτήρα για την ενότητά μας και για την αξιοπιστία μας στο να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έχουμε ενώπιον μας. Για μια ακόμα φορά αναφέρθηκε ότι το Καλίνιγκραντ είναι και αυτό μια άλλη βάση της ε, Ρωσίας και τώρα το Στρασβούργο μπορεί να κτύπηθει από πυράβλους από την Κρυμαία. Και από την Κρυμαία και από το Καλίνιγκρατ. Γι' αυτό υποστηρίζω την ιδέα. Χρειαζόμαστε καλύτερο συντονισμό με το ΝΑΤΟ και με τις ε, δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών και ένα κέριο στοιχείο για να μπορούμε να έχουμε ελπίδες για μια θετική αλλαγή στην Μαύρη Θάλασσα θα πρέπει να βασίζεται οποιαδήποτε τέτοια ελπίδα στο να έχουμε υπέρτερες ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις στην περιοχή. Σύμφωνο λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε <clears throat> ανοιχτοί για μακροχρόνια βελτίωση των σχέσεων μας με τη Ρωσία, αλλά στο βραχυπρόθεσμο <clears throat> και μεσοπρόθεσμο επίπεδο θα πρέπει να αλλάξουμε την οτροπία μας και να εστιάσουμε στις απαραίτητες αυτές αλλαγές που αφορούν πάρα πολύ τις χώρες της Μαύρης Θάλασσας, αλλά και όλους μας συνολικά. Ευχαριστώ κύριε Γκόμες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Πάσκου για την έκθεση που έρχεται αυτό το χρόνο. και υπογραμμίζει τα είδη των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε. Θα ήθελα να μας πει ο συνάδελφος πώς νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε. Γιατί αφενός υπογραμμίζει τη σημασία της υλοποίησης της δεύτερης συμφωνίας του Μίνσκ και την αποκλιμάκωση και άρα λύση με πολιτική συμφωνία και διαπραγμάτευση. Δεύτερον, όμως, Ξέρουμε ότι η συμφωνία του, η δεύτερη συμφωνία του Μίνσκ δεν αφορά το, την κρυμμέλα των πτώμα και δεύτερον, τρίτον μάλλον ποιο θα πληρώσει ή ποιος πληρώνει ήδη. Η ποιο πληρωνει ηδη η εναλλακτικη ποια θα ήταν λοιπόν. μια αποκλιμάκωση για την οποία έχει σημασία βέβαια η στρατιωτική παρουσία του ναυτικού στην περιοχή ή όχι. Και βέβαια πρέπει να κοιτάξουμε και τους ε, πολίτες, όχι μόνο τους Τατάρους που αναφέρθηκαν ήδη, αλλά τον ίδιο τον κόσμο στην Κρυμαία, πέραν των Τατάρων. Γιατί θέστηκαν πολλές ε, αναφορές από δημοσιογράφους τον τελευταίο καιρό και βλέπουμε ότι και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι πολλοί και εκτός των Τατάρων δεν είναι ευχαριστημένοι ότι την κατάσταση στην Κρυμαία τώρα μπορεί να λένε ότι αναγκάστηκαν να επιλέξουν μεταξύ δύο αλλά δεν είναι ικανοποιημένοι και δεν φαίνεται να βελτιώνει την κατάσταση του Νοτιού μάλιστα. Επομένως τι κάνουμε, περιμένουμε να εξελιχθεί η κατάσταση, ε, αναλαμβάνουμε κάποια δράση, δεν θέλουμε βέβαια να αντιδράσουμε κάποιο είδος πολέμου, αλλά πάντως σε καταστάσεις όπως αυτή που αντιμετωπίζουμε στην Ουκρανία, το κρίσιμο είναι ο κόσμος τι θέλει, τι ζητάει. Περαιτούμεθα ή κάνουμε μια προσπάθεια για αυτούς τους ανθρώπους στην Κρεμαία. Έχετε κάποια στρατηγική ενδεχομένω για να αντιληφθούν οι πολίτες τι είναι το καλύτερο. Ευχαριστώ κύριο Στάνακ. Υπήρχε ένα ενδιαφέρον άρθρο που διάβασα για αυτό το σημείο. Σήμερα το διάβασα στους Financial Times. Και έλεγε ότι υπάρχει ε, ένα πρόβλημα με τα τρόφιμα, περιθωρισμό το 8% κλείσαν τα σούπερ μάρκετ τα, τα, τα, ρωσικά και τους έφεραν από την Ρωσία ε, οι διατροφές. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι υπάρχει μεγάλη πίεση στον Πούτιν, ε, πολιτική πίεση σε σχέση με το ότι θα πρέπει τώρα εκεί πέρα να φτιάξει έναν ε, διάδρομο γιατί δεν μπορεί να δώσει αυτά που χρειάζονται οι πολίτες με, αυτό το εμπάργκο που έχει επιβάλει η Ουκρανία. Και ακριβώς βλέπουμε πώς έχουν τα πράγματα, γιατί χθε ο Πούτιν είπε στα μέσα ενημέρωση ότι άνετα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα πυρηνικά. Και το είχε πει στους διεθνείς ηγέτες ότι κινδυνεύουν Ρώσοι, πρόκειται περί ρωσικής επικράτειας και ότι ε, ανά πάσα στιγμή θα χρησιμοποιήσει τα πυρηνικά. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνος θεωρώ εγώ. Ε, είναι ακριβώς όπως έκανε η Σοβιτική, όπως έκανε και ο Μπρέσνιεφ Θυμάστε τότε που είχε εξαφανιστεί ο Μπρέσνιεφ, ε, εξαφανίστηκε για 10 μέρες, του ξεμφανίστηκε πάλι. Μιλάω όμως για πυρηνικά, πυρηνικό πόλεμο και, του, λέει ότι είναι δικαιωμά του, είναι δική του γη εκεί. Παρά το ότι 45% της περιοχής εκεί ε, δεν είναι Ρώσοι, είναι διάφορες μειονότητες και Ουκρανοί, ε, τους διώξανε, τους Οπότε βλέπετε πέρα πόσο μεγάλο πρόβλημα δημιουργήθηκε με τα ανθρώπινα δικαιώματα και νομίζω ότι ε, ε, Ιαν ε, είσαι πολύ γενναιόδωρος εκεί στην εκλογή παράγραφο G που και την Τουρκία και το διάβασα και το ξαναδιάβασα εκεί το ότι δηλαδή επιδεικνύει αλληλεγγύη, πολύ μεγάλη αλληλεγγύη προς το Αζερμπαϊτζάν, προς τους τουρκογενείς που πέφτουν στο Ναγκόρνο Καραμπάχ. Τώρα όμως τι γίνεται με τους Τάταρους που υποφέρουν τόσους ε, αιώνες. Θυμηθείτε τι έγινε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, είναι στην ε, σφαίρα επιρροής της και είδατε ότι υπήρξε προσέγγιση με τον ε, Ερντογάν γιατί πρόκειται μεταξύ δύο ουσιαστικά δικτατόρων. Μην το ξεχνούμε αυτό. Επίσης κάτι άλλο που διάβασα στους Financial Times σήμερα ότι ο Σεύκοβιτς και ο που είναι η αρμόδια επίτροπη και ο δεύτερος για τον, ε, για τον ανταγωνισμό. Τώρα θα, θα, θα λάβουν μέτρα κατά της Gazprom λόγω της προσάρτησης της Κρυμαίας. Ε, είχαν διακόψει τότε που είναι δηλαδή οι προσάρτηση και τώρα θα ξαναρχίσουν και η Gazprom επειδή ε, εφαρμόζει κάποιες καταπλεονεστικές πρακτικές πρόκειται να υποστεί μεγάλο πρόστιμο και αυτό αφορά και τις ε, βαλτικές χώρες. Να, τι μπορούμε εμείς να χρησιμοποιήσουμε ως δημοκράτες, ως οικονομικά όπλα για όλα αυτά τα οποία έκανε η Ρωσία και κράτησε πάρα πολύ αυτό το οποίο έκανε. Πρέπει να μας προβληματίσει αυτό σε σχέση με την έκθεση. Επίσης αναφέρθηκε το θέμα του Καλίνιγκραντ και στα πλαίσια των κυρώσεων θα πρέπει να σταματήσει αυτό το καθεστώς το οποίο χωρίθηκε στους Ρώσους για την ε, διέλευση. Ελεύθερη διέλευση, ούτε βίζες ούτε τίποτα. Αυτό το εκχωρήσαμε στους Ρώσους και μπορούμε να το πάρουμε πίσω. Να το κάνουν τα, τα όμορα κράτη. Στα πλαίσια των κυρώσεων. Επίσης, είσαι πάρα πολύ κοινάδος όσον αφορά την Τουρκία. Εκεί που λες για το Ισλαμικό κράτος. Αλλά νομίζω ότι όλα τα στοιχεία, τότε που απελευθέρωσαν εκείνο τον ε, ναό κοντά στο κομπάνι στην Βόρεια Συρία, τότε υπήρξε αυτή η εκεχηρία και δεν έπεσε ούτε ντουφεκιά τότε που πήγε το Ισλαμικό κράτος και και κάποιους Τούρκους. Δηλαδή, με, με την τάση με το Ισλαμικό κράτος, έχει ανοιχτό διάβλο επικοινωνία η Τουρκία. Λοιπόν, στους παντούς είναι απελευθέρωση των ομήρων πριν από λίγο καιρό. Πώς όμως θα θεωρήσουμε ότι είναι εχθροί. Άρα να το δούμε αυτό. πώ θα χτενίσουμε το κείμενο με κάποια τροπολογία. Γιατί θα πρέπει να φέρουμε και στον ε, Πούτιν, ο οποίο ήταν έτοιμο να χρησιμοποιήσει πυρηνικά γιατί θεωρείται είναι έδαφο τη Ρωσία και ότι ο λαό ο ρωσικό, κινδυνεύει από το Κίεβο. πρόεδρο. Και θα τον ευχαριστούμε κύριος Φραντζολίτσα. First uh, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να συγχαρώ τον εισηγητή πρώτα απ' όλα για την πληρότητα της έκθεσής του. Μόνο μερικά σχόλια σε σχέση με την κατάσταση στη Μαύρη Θάλασσα. Αν δείτε τη χερσόνησο της Κρυμαίας, έχει το μέγεθος του Βελγίου σχεδόν. Ε. λίγο λιγότερο από το Βέλγιο. Είναι σαν ένα μεγάλο αεροπλανοφόρο στη Μαύρη Θάλασσα. Όποιος ελέγχει την Κρυμαία ελέγχει και τη Μαύρη Θάλασσα. Από τη στιγμή λοιπόν που η Ρωσία έχει καταλάβει την Κρυμαία και έχει ενισχύσει τη στρατιωτική της παρουσία με τους πυράβλους Ισκεντέρ είναι πολύ πιο ισχυρή η παρουσία της και φυσικά μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτούς τους πυράβλους και με πυρηνικές κεφαλές ακόμα. Αν δούμε την κατάσταση στην Ανατολική Ουκρανία. Νομίζω ότι απλώς έχουμε μια σύντομη ανάπαυλα. Η Ρωσία δεν θα σταματήσει. Ελέγχουν τώρα την Ανατολική Ουκρανία. Έχουν στην κατοχή τους την Νότια Ουκρανία και την ε, Κρυμαία και έχουν και μια παρουσία στη Δυτική Ουκρανία με την υπερνηστερία. Η Ουκρανία λοιπόν βρίσκεται σε ένα κλειό και όπως ελέγχεται από πολλούς η Ρωσία ετοιμάζεται να καταλάβει το σύνορο της Ουκρανίας. Κατά την άποψή μου η απάντηση της δύση και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επιθετικότητα αυτή της Ρωσίας γιατί δεν ε, πιστεύω ότι οι αποσχιστικές δυνάμεις είναι αυτόνομες στην Ανατολική Ουκρανία αυτόνομες από τη Ρωσία, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ήταν πάρα πολύ ήπια, ήταν πολύ αδύναμη ουσιαστικά η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη ρωσική επιθετικότητα και σε όλη την ιστορία της Ευρώπης οι παρεμβάσεις της Ρωσίας στα Βαλκάνια, στις Βαλτικές χώρες έχουν καταδείξει ότι όταν ε, διαβουλεύεται κανείς με τη Ρωσία σε διπλωματικό επίπεδο, η Ρωσία βγάζει το συμπέρασμα ότι είμαστε αδύναμοι. Μόνο τη βία καταλαβαίνουν, μόνο τη δύναμη. Κάπου πρέπει να τη σταματήσουμε. Γιατί αλλιώς κάποιες από τις χώρες μας μπορεί να κινδυνεύσουν να χρειαστεί να πολεμήσουν τη Δυτική Ουκρανία για να υπερασπιστούν τα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης. Δεν θέλω να επικαλεστώ την αποκάλυψη του Ιωάννη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Αλλά νομίζω ότι ορισμένοι λαμβάνουν υπόψη τα θέματα αυτά με πραγματικά υπερβολικά ήπιο τρόπο, με άσπρα γάντια, πηγαίνουν στη Ρωσία για να έχουν νέες οικονομικές συμφωνίες προς όφελόν τους. Αυτό δεν είναι μια κοινή όμως πολιτική άμυνας και ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ρωσία ήταν έτοιμη να κάνει ασκήσεις αεροπονικών δυνάμεων μαζί με την Σερβία το Σεπτέμβριο στα σύνορα της Ρουμανίας σε, με ενόπλων ε, δυνάμεων της αεροπορίας τους. Θα πρέπει και εδώ να εκφράσουμε λοιπόν την ανησυχία μας ήδη να σε αυτή την έκθεση λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό είναι μια πρόσθετη <clears throat> πρόκληση ε, έναντι των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε στη Σερβία, η οποία θέλει να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι θα πρέπει να συμμορφωθεί με την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχει βεβαιωτή πολιτική, παρά μόνο στα χαρτιά. Και γι' αυτό η Ρωσία μπορεί να εκμεταλλεύεται τόσο πολύ αυτές τις ευκαιρίες που της δίνουμε. Θα πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν πώς θα αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες που μας δημιουργεί η πράξη αυτή της σερβικής κυβέρνησης σε σχέση με τις κοινέ αυτές ασκήσεις σε σερβικό έδαφος. Και ξέρετε ότι η σερβική αεροπορία, <clears throat> πολεμική αεροπορία, εκπαιδεύεται και εφοδιάζεται από την Ρωσία. Λυπάμαι πάρα πολύ κυρίες και κύριοι που δυστυχώς οι χώρες της δύση και η Ευρωπαϊκή Ένωση κρατούν μια αμυντική στάση έναντι των ρωσικών προκλήσεων και στρατιωτικών δράσεων στην Ουκρανία και αλλού. Στον ε, κυβερνόχωρο επίσης, έναντι του υβριδικού πολέμου που ασκεί η Ρωσία και των άλλων προκλήσεων όπως είναι οι συμφωνίες της Ρωσίας με πολιτικά κόμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της επιδότησης που δίνει η Ρωσία σε κόμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έχετε δει όλο αυτό, το είδατε και στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν ο κύριος Πούτιν παίρνει υποστήριξη από διάφορους βουλευτές που ξέρετε σε ποιο κόμμα ανήκουν. Είναι καιρός λοιπόν κυρίες και κύριοι να υψώσουμε το ανάστημά μας και να έχουμε μια ισχυρή θέση να της Ρωσίας. Ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φουντζούλητσα. Ο κύριος Γκάλερ τώρα για δικό του λογαριασμό και στα αγγλικά. Ευχαριστώ. Μερικές παρατηρήσεις, μερικές ε, υποδείξεις. Μια και είμαστε στον, στην ΟΑΣΕ και έχει και λειτουργικό ρόλο, δεν μπορούμε να κάνουμε μια αναφορά σε αυτό, ζητώντας τη Ρωσία να δώσει πρόσβαση σε όλους, ε, σε ολόκληρη την επικράτεια, όπου χρειάζεται, εν πάση περιπτώσει, και γιατί όχι και στην Κρυμαία. Είναι μέλος της ΟΑΣΕ η Ρωσία και ως εκ τούτου θα πρέπει σήμερα με εμπιστοσύνη να συνεργάζεται με την οργάνωση αυτή. Εάν θέλει η Βάση και κάποια από τα κάποια της να μεταβεί και να κάνει κάποια πράγματα γνωμοσύνη στην Κρυμαία, πρέπει να επιτραπεί. Το ίδιο και με το Συμβουλίο της Ευρώπης, ακόμη περισσότερο μάλιστα, καθώς ε, έχουμε να κάνουμε με ανθρώπινα δικαιώματα. ζητάει την πρόσβαση στην Κρυμαία. Σε τελευταία ανάλυση η Κρυμαία είτε ανήκει στην Κρυμαία όπως εμείς θεωρούμε, είτε στη Ρωσία όπως θεωρούν οι Ρώσοι, είναι κομμάτι του Συμβουλίου της Ευρώπης. Άρα θα πρέπει οι Ρώσοι να επιτρέψουν σε μια αντιπροσωπεία ε, μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης να πάνε να εξετάσουν την κατάσταση και να δουν ποια είναι η κατάσταση με τη διαφάνεια και βέβαια την ασφάλεια. Και επίσης έχει ε, δηλώσει πως είναι ανυπόστατη η συμφωνία το μνημόνιο καλύτερα της Βουδαπέστης η Ρωσία. Και αν όχι, οι λοιποί υπογράφοντες Βρετανία, Ηνωμένε Πολιτείε, Ουκρανία δεν θα μπορούσαν να απαιτήσουν δυνάμει του μνημονίου αυτού του, της Βουδαπέστης να γίνει μια συνεδρίαση για τα θέματα αυτά που προβληματίζουν. Δεν θα έπρεπε λοιπόν πρώτα να αναφερθούμε στο μνημόνιο της ε, Βουδαπέστης. Και να στήσουμε από τα άλλα συμβαλόμενα μέρη να καλέσουν τη Ρωσία να συνομιλήσει για θέματα που έχουν να κάνουν με την εδαφική αικαιρότητα της Ουκρανίας. Ευχαριστώ, λέει και πρόεδρος. Υπάρχει κάποιο άλλο ο οποίο θέλει να λάβει το λόγο. Όχι, οπότε θα ξαναδώσω το λόγο στον κύριο Πάσκου. Σα ευχαριστώ πολύ. Υπήρξαν μερικέ πολύ καλέ προτάσει, οι οποίε θα βρουν αντίκρισμα και στην έκθεσή μου. Το πρόβλημά μου είναι ότι υπάρχει πάντα ο περιορισμό των αριθμών των λέξεων. Άμα βάλετε μια λέξη, πρέπει να βγάλετε μια άλλη. Πολλά πράγματα λοιπόν τα οποία εγώ ήθελα να πω ή να επεκταθώ σε αυτά ή ήμουν υποχρεωμένος να τα πω πιο συνοπτικά ή να τα αφαιρέσω. Αλλά σίγουρα τα μέλη μπορούν να δημιουργήσουν και κάποιο περιθώριο περαιτέρω με τις τροπολογίες τους. Συμφωνώ λοιπόν ότι πρέπει να δώσουμε περισσότερη προσοχή στα πυρηνικά όπλα. Ο κύριος Πούτιν είπε ότι θα μπορούσε να αυξήσει το επίπεδο ετοιμότητας του πυρηνικού προστασίου της Ρωσίας. Βέβαια, κάποιοι άλλοι λένε ότι η Ρωσία έχει κάθε δικαίωμα να έχει πυρηνικά όπλα στην Κρυμαία. Και υπάρχουν και δηλώσεις των Ρώσων αξιωματούχων από την άποψη αυτή. Πρέπει λοιπόν να ληφθεί υπόψη και το θέμα του πυρηνικού οπλοστασίου. οι Τατάροι και η Άννα ανέφερε ότι δεν πρέπει να αφήσουμε και τον υπόλοιπο πληθυσμό. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε μονάχα τους Τατάρους. Όχι. Αλλά είναι οι Ουκρανοί οι οποίοι βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση. Είναι το δικό τους ε, έδαφος. Δεν μπορούμε να δώσουμε στους Ουκρανούς κάτι το οποίο δεν διεκδικούν οι ίδιοι. Πρέπει να λάβουμε υπόψη όμως και τον υπόλοιπο πληθυσμό. Τα επιχειρήματα του Προύτιν είναι ότι η νομιμότητα των ενεργειών του βασίζεται στο ότι έχουμε στείλει στην Κρυμαία εκπροσώπους των δυνάμεων πληροφοριών αλλά ήταν κάτω από το, την οροφή των 20.000 που μπορούν να έχουν στη Σεβαστούπολη, επομένως αυτό είναι νόμιμο. Αλλά η προσάρτηση, πού τη βάζουμε την προσάρτηση. Είπε ότι βασίζεται σε ένα δημοψήφισμα που έγινε στην Κρυμαία, δηλαδή επί τη βάση θέλησης του πληθυσμού. Είμαι ο τελευταίος ο οποίος θα αναφερθεί σε άλλες περιπτώσεις ε, στην ιστορία όπου ο πληθυσμός αποφάσισε ε, με κάποιο δημοψήφισμα το οποίο μπορεί να ήταν ε, αμφισβητήσιμης ε, Αλλά δεν μπορούμε να θεωρήσουμε νόμιμο αυτό το οποίο έχει γίνει. Πρέπει να σκεφτούμε περισσότερο και την γεωργία, τι έχει γίνει και τι θα γίνει με την γεωργία στο μέλλον. Γιατί αν δούμε τις χώρες αυτές, τι βλέπετε. Βλέπετε ότι μας είχαν ζητήσει το 2008 στο Βουκουρέστι ένα σχέδιο δράσης που δεν το δεχτήκαμε. Και τους είχαμε υποσχεθεί να γίνουν ακόμα και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είπε ο Πούτιν ότι ήθελε να εμποδίσει κάτι τέτοιο. Αποφάσισε λοιπόν να ουσιαστικά να σακατέψει αυτές τις χώρες για να μην είναι επιλέξιμες ως δυνητικά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όταν τώρα ζητούν τη βοήθειά μας, τους λέμε δεν είσαστε μέλη του ΝΑΤΟ, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτά είναι τα ηθικά και νομικά διλήμματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε αυτήν την περίπτωση. Φυσικά πρέπει να εξετάσουμε και την περίπτωση της Gazprom, την οικονομική πτυχή των θεμάτων αυτών. Από ό,τι ξέρω η Ροσμέτ έχει αγοράσει από τη Γεωργία το εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερού στο Ερτοπότ. Πρέπει να το ελέγξουμε αυτό κατά πόσο ισχύει ή όχι. Αλλά και εκεί παίζεται το παιχνίδι με το Ισλαμικό κράτος. Ναι, βεβαίως, το μόνο πρόβλημα το οποίο εγώ θέλω να υπογραμμίσω είναι το ότι η Τουρκία, ό,τι πολιτικό παιχνίδι και να παίζει προς το παρόν, παραμένουν κέρια χώρα στον αγώνα κατά του Νταές, Ισλαμικού κράτους. Αν θα χρησιμοποιήσουν όλη τη δύναμή τους οι Τούρκοι, αυτό εξαρτάται από την πόση πρόσβαση θα μας επιτρέψουν να έχουμε στο πλήρες δυναμικό τους. Δεν ήμουν γενναιόδωρος, θέλω απλώς να υπενθυμίσω αυτό το γεγονός και να σας πω ότι έχουμε δύο απειλές εδώ στη Μαύρη Θάλασσα. Έχουμε απειλές τύπου Ισλαμικού κράτους στο Νότο και στην Τουρκία και έχουμε την παραδοσιακή απειλή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την Κρυμαία και παίζουν όλες αυτές οι απειλές στον ίδιο περίπου ε, γεωγραφικό χώρο. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Τάραντ, ο οποίος είπε να συνεχίσουμε τις έρευνές μας στα τμήματα αυτά τα οποία δεν είναι υπό τον έλεγχο της ε, κυβέρνησης της ε, Ουκρανίας. Αλλά θυμάμαι το αστείο με το αρμενικό ράδιο όταν ζήτησε κάποιος, ρώτησε κάποιος στο ράδιο Γερεβάν πόσο παίρνει ένας ε, Ρώσος εργαζόμενος. Και η απάντηση ήταν «Μα εσείς δεν σκοτώνετε τους μαύρους στις Ηνωμένες Πολιτείες». Η απάντηση στον Αμερικανό αυτό δημοσιογράφο. Βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα χώρο όπου εγώ θέλω να ενοχληθώ, ό,τι και να πείτε θα με ενοχλήσει αυτό που μου λέτε και όσο μου τα λέτε περισσότερο, τόσο περισσότερο ενοχλούμε τα μηνύματα λοιπόν τα οποία στέλνουμε και η προσπάθεια να μην ενοχλούμε τους Ρώσους γιατί θα κάνουν κάτι κακό, αυτό δεν νομίζω ότι αυτό είναι η λύση. Ήδη έχουν κάνει κάτι το αρνητικό και το παράνομο χωρίς εμείς να τους προκαλέσουμε. Αλλά συμφωνώ και εδώ θα κλείσω ότι έχουμε ένα πρόβλημα γιατί το Μίνσκ 2 αναφέρεται στην περιοχή του Λουγκάνσκ και του Ντονμπάς, αλλά δεν λέει τίποτα για την Κρυμαία προς το παρόν. Έχουμε λοιπόν τις κυρώσεις, έχουμε την μη αναγνώριση, η οποία θα εξακολουθήσει να ισχύει, αλλά συγχρόνως, τέλος κάτω στα θέματα θα παραμείνουν στην Κρυμαία και θα κάνουμε ό,τι θέλουν στην Ουκρανία. Περίπου. Δεν έχουμε λοιπόν κάποια ορατή λύση. Εκτός αν κάνουμε κάποια δυναμική ενέργεια ή κάτι το εντυπωσιακό που κανείς δεν ξέρει τι θα μπορούσε να είναι. Όταν μιλάμε με μια ηγεσία η οποία μιλάει για πυρηνικές απειλές τώρα και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το σκεφτούμε. Ελπίζω λοιπόν ότι θα επανέλθουμε και εγώ σας υπόσχομαι θα λάβω υπόψη πάρα πολύ σοβαρά όλα αυτά που είπατε. Προσπάθησα να δώσω απαντήσεις σε ορισμένα από αυτά. Θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι για τις ε, προτάσεις σας και τις συστάσεις σας και θα προσπαθήσω να βελτιώσω την έκθεση αυτή όσο μπορώ περισσότερο. Ευχαριστώ. I like to... Ευχαριστώ. Ήθελα να προσθέσω ένα-δύο σημεία οπωσδήποτε τη δεύτερη συμφωνία του Μίνσκ και την Κρυμαία. Την εποχή του Μεϊντάν πολλοί ήταν οι Ρωσόφωνοι που δήλωναν ότι δεν θα δεχόντουσαν οποιαδήποτε εμπλοκή και παρουσία της Ρωσίας στην επικράτεια. Ήταν άλλωστε και η πρώτη απόφαση του Γιαννούκοβιτ αυτή από την ανάληψη της εξουσίας να επεκτείνει την διάρκεια της συμφωνίας για την Σεβαστούπολη και την παρουσία του στόλου. Πάντως οπωσδήποτε πρέπει να υπαλληθεύσουμε αυτά που λέτε και οπωσδήποτε πρέπει να κοιτάξουμε για το πότε ειδικά και μετά την κατάρρευση της ε, κυβέρνησης του Αλασάνιας, του κόμματος Αλασάνιας. Έγιναν κάποιες σιωπηλές αλλαγές προσώπων ο Υπουργό Άμυνα που είναι υπεύθυνο και για θέματα του ΝΑΤΟ προέρχεται από το κόμμα Πουτσενάτα. Άρα υπάρχει ζήτημα αύξηση τη σφαίρα επιρροή. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι προθεσμία για την καταστροπολογιών έχουμε έως τις 23 Μαρτίου, 12 το μεσημέρι. Θα ξανασυστήσουμε την πρόταση 16 Απριλίου. Η ψηφοφορία θα γίνει στην ΑΦΕΤ φυσικά. Για αύριο υπενθυμίζω στους συντονιστές ότι έχουμε ένα διευρυμένο προεδρείο στις 9 και αρχίζουμε στις 10 τη συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ.